Καλημέρα σε όλους σας. Αν δεν έχετε αντίρρηση θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής. Καταρχήν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με κάποια σχόλια του Προέδρου. Πολλές πολιτικές ομάδες ε, ζήτησαν και συμφώνησαν όλες ως προς την ε, ψηφοφορία της έκθεσης στη Βέσο για την ΚΟΑ και Χάρτλουγκ για τον κανονισμό 2371 ε, του 2002 να αναβληθούν οι, οι ψηφοφορίες αυτών των δύο εκθέσεων για τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας του Ιουνίου. Οπότε το σημείο 14, την έκθεση Μιράντα δηλαδή για την ειδική έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου θα την εξετάσουμε Στι 10 και 4, με το που θα τελειώσουμε την ψηφοφορία, τη μοναδική ψηφοφορία που έχουμε για την Πέμπτη. Και το σημείο 9, έκθεση Φεραίρα δηλαδή για τη μικρή κλίμακα ελία και παραδοσιακή ελία θα την συζητήσουμε την Πέμπτη και όχι σήμερα ως τελευταίο σημείο. Την Πέμπτη 11 η ώρα, αύριο 11 η ώρα το πρωί. Μια άλλη αλλαγή αφορά το σημείο 15, το Σολομό της Βαλτικής, την έκθεση Γκρομπάρτσικ που θα γίνει σημείο 21. Ενώ το 21 θα συζητηθεί ως 15ο. Θα γίνει μια αντιστροφή των σημείων 15 και 21 στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή για αύριο. Αν δεν έχετε αντίρρηση, εγκρίνουμε με τις αλλαγές αυτές στην ημερήσια διάταξή μας. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών της 23ης και 24ης Απριλίου. Θα θεωρηθούν εγκεκριμένα αν δεν υποβληθούν στη διάρκεια της συνεδρίασής μας, της σημερινή ε, διορθώσει ή αντιρρήσεις. Ανακοινώσεις του Προέδρου δεν υπάρχουν και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4, την ακρόαση δηλαδή, για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, ΕΤΘΑ. Για το πρώτο αυτό σημείο θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τους ε, εμπειρογνώμονές μας, τους προσκεκλημένους σε αυτή τη συνεδρίαση γιατί θα ξεκινήσουμε αμέσω ε, την δημόσια κρόση. Του ευχαριστώ θερμά του καλεσμένου που ήρθαν για να μα μιλήσουν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αιλίες. Θα μα αναλύσει τα προβλήματα του υπάρχοντο ταμείου και τι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τι δυσκολίε του μέλλοντος. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η δημόσια κρόση και πολύ επίκαιρη. Είχαμε και άλλε ακρόασει για διάφορου άλλου κανονισμού και θέματα που μα απασχολούν. Αυτή η δημόσια κρόση, επαναλαμβάνω, διοργανώνεται σε μια κέρια και πολύ επίκαιρη στιγμή. Το νέο ταμείο περιλαμβάνει πολύ θετικά σημεία, γιατί στόχο έχει μια βιώσιμη αλληλιακή υδατοκαλλιέργεια, αλλά περιλαμβάνει και κάποια αρνητικά σημεία, κάποιες αδυναμίες που φαντάζομαι θα αναδειχθούν στη διάρκεια της σημερινής δημόσιας ακρόασης, προκειμένου να βελτιώσουμε στο μέτρο του δυνατού τη λειτουργία αυτού του νέου ταμείου. Μερικά διαδικαστικά, οργανωτικά για τη δημόσια κρόση. Ως συνήθω, θα έχουμε δύο πάνελ. Το πρώτο αφορά την ε, εμπειρία και τις δυσκολίες από την ε, διαχείριση του ισχύοντος Ταμείου Αλίας και προτάσεις για τη διαχείριση του νέου Ταμείου Αλίας. Ο κάθε καλεσμένος έχει γύρω στα 10-13 λεπτά για να μείνει λίγος χρόνος και για συζήτηση αργότερα. Πρώτα θα μιλήσει ο κ. Σερμίδα Τραστό, ο Γενικός ε, Διευθυντής ε, ε, για την Αλία του Υπουργείου Ιαλίας. Μετά η κυρία Γιαντζέβα Παλασόβα, Γενική Διευθύντρια του, της Εθνικής, της Εθνικής Οργάνωσης Αλίας της Ισπανίας. Και μετά ο κ. Κούκα, που είναι σύμβουλος του Υπουργείου του Φιλανδικού Υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομείας. Θα γίνει μια συζήτηση και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Πρώτα θα δώσω όμως το λόγο στον κύριο Ελέν Καντέκ, τον συνάδελφο Καντέκ, που είναι και ο εισηγητής της πρότασης κανονισμού για το νέο Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Ευχαριστώ θερμά όλους. Κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μια καθοριστική στιγμή, ορόσημο για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική, οπότε το ταμείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί σε αυτή την ακρόαση. Θα ήθελα εδώ να έχουμε την ευκαιρία, στο νομοθετικό μα ρόλο, να ακούσουμε του εκπροσώπου του τομέα αυτού και να τροφοδοτήσουμε και τη δική μα συζήτηση με τι δικέ του εμπειρίε. Πρόεδρε, ευχαριστώ του προσκεκλημένου μα που προσήλθαν. Δεν έχουν φτάσει βέβαια όλοι. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα φτάσουν. Και σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε τα τρία σημαντικότερα σημεία της μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική, τον ε, βασικό κανονισμό, την κοινή οργάνωση αγοράς ε, με εισηγητή τον κύριο Στίβενσον και το ταμείο το οποίο έχω αναλάβει εγώ ως εισηγητής το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλία έχει αλλάξει πλέον ονομασία και ονομάζεται Ευρωπαϊκό Ταμείο για, τη θάλα, για τα θαλάσσια ζητήματα και την αλία. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από την τροπή που θα πάρει ο βασικός κανονισμός εδώ, αλλά εγώ μιλώ για μια ουσιαστική τροποποίηση του κανονισμού αυτή στην έκθεσή μου. Διότι ιδάλλως θα έχουμε ένα εργαλείο που θα συνοδεύει την επαγγελματική αλλαγή, την ε, ε, αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης των αλλιών του τομέα και την ε, στήριξή τους εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο που δεν είναι ευκταίο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε σε πρώτη προτεραιότητα και αυτό προτείνω στην εκθεσή μου την προστασία των αποθεμάτων. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε μαζί με την Επιτροπή τις πλεονάζουσες δυνατότητες του στόλου ακόμη και σαν ορισμένα αλληλευτικά αποθέματα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα οριστεί η δυνατότητα και η πλεονάζουσα δυνατότητα. Θα πρέπει να συζητηθεί η διαπίστωση αυτή, διότι η ικανότητα ακόμα δεν έχει ζητηθεί επαρκώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δύσκολο να παληθευτεί. Ορισμένες περιοχές έχουν αλληλευτικές δυνατότητες πολύ ε, μεγάλες σε σχέση με το τι δυνατότητες διαθέτουν στα χέρια τους και θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα ορίσουμε και τις ζώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το βασικό κανονισμό και την πρόβλεψη ε, μεταβιβάσιμων αδειών αλίας. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να καλύπτει και την ε, μικρή κλίμακα αλλία και την παραδοσιακή και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη ως πρόταση. Πιστεύω ότι εδώ συμφωνούν πολλοί συνάδελφοι. Η αλλία αυτή, η μικρή κλίμακα και παραδοσιακή ε, πρέπει να διαφυλαχθεί στο μέλλον στην Ευρώπη. Διότι 30% των αλληλευτικών προϊόντων που καταναλώνουμε προέρχονται από την Ιδωτοκαλλιέργεια και την αλληλεία αυτή. Πρέπει λοιπόν να προστατέψουμε και τα αποθέματά μα και να σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπερβολικά πολλού κανόνε, περισσότερο από κάθε άλλο μέρο στον κόσμο. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι συμβατά όλα αυτά με τον βασικό κανονισμό βέβαια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι γυράσκει ο Ευρωπαϊκό Στόλο και εδώ, με πηγή την Eurostat, πρέπει να δούμε κατά πόσον, ε, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, γίνονται σεβαστές οι ανάγκες ασφάλειας και κατά πόσον μπορούμε να ανανεώσουμε το στόλο βάσει αυστηρών προδιαγραφών. Θα πρέπει να ε, ενθαρρύνουμε την ε, αλία με καλύτερες μεθόδους και όχι τον περιορισμό σε ποσότητα. Υπό προϋποθέσεις. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό των σκαφών και αυτό υπό συγκεκριμένου όρου. Να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια, την κατανάλωση ενέργειας κατά τρόπο σημαντικό τη ρήπανση και να προωθήσουμε επιλεκτικότερες και προηγμένες, προηγμένα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται. Εδώ Ξέρουμε ότι κάποιες από τις προτάσεις δεν είναι δυνατόν να ε, εφαρμοστούν σε σχέση με τη διάλυση των σκαφών. Εγενεόδορες προτάσεις κάνει η Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να δούμε και το ρεαλιστικό με μια σταδιακή ε, προσαρμογή τους. Εδώ για τη διάλυση σκαφών θα πρέπει να δούμε τι είναι συμφερότερο. Να διατηρηθούν κάποια σκάφη στην, ε, στον τομέα ή να αντικατασταθούν εφόσον είναι απαρχαιωμένα. Όμως, θα πρέπει να αναζητήσουμε σκάφη ενεργειακά αποδοτικότερα, ασφαλέστερα και πιο επιλεκτικά. Ίσως και μικρότερης ισχύω. Θα πρέπει πάντως να δούμε πόσο μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την ε, απόδοση των σκαφών. Επίσης, εδώ δεν φαίνεται να προβλέπεται στήριξη για τους επαγγελματίες της αλίας που προσωρινά έχουν πάψει τις δραστηριότητε τους σε περίπτωση μεγάλων οικολογικών ατυχημάτων ή δυσμενών κλιματολογικών συνθήκων. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν εδώ κάποιοι κανόνε για να προστατεύονται αυτοί οι επαγγελματίε που προσωρινά έχουν πάψει τι δραστηριότητέ του. Έπειτα, η αύξηση των τιμών των καυσίμων βαρύνει ιδιαίτερω τι ε, μικρέ ε, μονάδε αλεία. Το ζούμε αυτό στι παράκτητε περιοχέ πολλών χωρών. Θα ήθελα λοιπόν να προβλέπεται ένας μηχανισμός προσωρινής ισχύω για αντιστάθμιση του υπερβολικού αυτού κόστου, ώστε να μπορούν οι αλλοί να διατηρούν την δραστηριότητά του σε περίπτωση που έχει αυξηθεί υπερβολικά η τιμή του καυσίμου, των καυσίμων του. Είχαμε προβλέψει κάποια κονδύλια 30.000 ευρώ ντεμίνιμη εξελαχίστων στα, σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να προβλέψει λοιπόν κανόνε ισότι, κανόνες ισότιμους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο γίνονται σεβαστοί οι κανόνες της ε, κοινοτικής πολιτικής αλίας και εδώ καλωσερίζω τις φιλόδοξες προτάσεις της Ευρωπαϊκής σχετικά με το θέμα αυτό. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μια προσπάθεια για να υπολογίσουμε τα βιώσιμα επίπεδα για όλα τα αποθέματα που είναι αντικείμενα εμπορία. Αυτό είναι σημαντική προτεραιότητα. Θα πρέπει επίσης να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει συνεργασία των επαγγελματιών με επιστημονικέ επιτροπέ, για να συλλέγονται δεδομένα, να υπάρχουν ε, συγκεκριμένε μελέτε και να καταρτίζονται και οι καλύτερε πρακτικέ. Η πρόταση τη Επιτροπή έχει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο κεφάλαιο και για την ε, καλλιέργεια τη υδατοκαλλιέργεια, για την στήριξή τη μάλλον. Εδώ θα πρέπει να ενθαρρύνουμε του ε, διάφορου επενδυτέ να ασχοληθούν με τον τομέα αυτό. Καλωσορίζω ορίζω λοιπόν τι προτάσει τη Επιτροπή σχετικά. Σε σχέση με την ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπολογίζει ένα κονδύλι 430.000 ευρώ μέχρι το 2020. Τετραπλασιάζει δηλαδή τον προπολογισμό τη πολιτική αυτή στα πλαίσια του Ταμείου. Θα πρέπει να δούμε αν τα κονδύλια αυτά είναι επαρκή για να έχουμε σωστή διακυβέρνηση στη θάλασσα και την τον καλό έλεγχο του θαλάσσιου χώρου. Αλλά αυτά να μην γίνουν ει βάρο τη αλληλευτική πολιτική και τη θεατοκαλλιέργεια. Θα πρέπει λοιπόν να αναλυθεί λεπτομερώ η ε, δημοσιονομική πρόταση και να βρούμε έναν κανονισμό που να μπορεί να στηρίξει τι ε, φιλοδοξίε αυτέ. Συνάδελφοι, φίλοι, ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλία όντω θέλουμε να είναι φιλόδοξο για να εξασφαλίσουμε και το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Αλία. Το Ταμείο αυτό δεν θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο για να αλλάζουν επαγγελματική δραστηριότητα ή αλίε εφόσον χρειάζεται, κάτι που προτείνει η Επιτροπή, αλλά να του επιτρέπει να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται σε καλέ συνθήκε. Να είναι ένα πλαίσιο για μια βιώσιμη αλία. Ε, κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν η εισήγησή μου. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους προσκεκλισμένους μας, που και πάλι θέλω να ευχαριστήσω για την προσέλευσή Νομίζω θα είναι σημαντική η μαρτυρία τους για να εμπλουτιστούν οι εργασίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καντέκ. Πολύ χρήσιμες αυτές οι εξηγήσει, γιατί θέλετε ένα φιλόδοξο ταμείο. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινή επιθυμία. Παρόλο που για μερικά από τα επιμέρους θέματα υπάρχουν διαφωνίες. Περνάμε τώρα στη δημόσια κρόση και δίνουμε το λόγο στον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Αντρέ Ερμίδα Τραστόη, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Ελίας του Ισπανικού Υπουργείου ε, Γεωργίας, ε, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Παρακαλώ να μην ξεπεράσετε το χρόνο σας, τα 13 περίπου λεπτά, για να μας μείνει χρόνος ε, για τη συζήτηση. Θα ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων γιατί θα λείψω λίγο, έχω μια ενηλυμένη υποχρέωση, αφήνω στα χέρια του Αντιπρόεδρου Στίβενσον την διεξαγωγή της ε, δημόσια κράτησης προς το παρόν. Κύριε Ερμίδα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μου δίνει την ευκαιρία να σας ε, παρουσιάσω την εμπειρία της Ισπανίας στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας, του ΕΤΑ, τις δυσκολίες ε, στην εφαρμογή του που αντιμετωπίσαμε, ώστε να αποφευθούν ε, στο νέο Ταμείο Αλίας, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, το ΕΤΘΑ. Ελπίζω ότι η εμπειρία μας από τη διαχείριση του 26,29% του συνόλου των κονδυλίων του Ταμείου Αλίας 2007-2013 θα είναι ενδιαφέρουσα για να βελτιωθεί η διαχείριση και του νέου ΕΤΘΑ. Ο κανονισμός του ΕΤΑ ε, στηρίζεται σε μια δομή προγραμματισμού που φαίνεται λογική. Απαιτείται ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, σχέδιο με τις βασικές γραμμές πολιτικής δράσης στις οποίες θα στηρίζονται τα μεταγενέστερα έγγραφα προγραμματισμού. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που περιλαμβάνει κάποιες διαρθρωτικές δράσεις καθώς και μια οργανωτική διάρθρωση που θα πρέπει να ε, εγγυάται το, την ευόδοση των δράσεων. Σε μεταγενέστερη φάση απαιτείται από τα κράτη-μέλη η εκπόνηση του εγγράφου διαχείρισης και ελέγχου. Εκεί περιλαμβάνονται αναλυτικά οι διοικητικές διαδικασίες για τη διαχείριση των ενισχύσεων και μάλιστα εγκρίνεται από την ε, αρχή ελέγχου. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα κριτήρια επιλογής των σχεδίων που ε, εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε κράτους μέλους. Η εκπόνηση αυτών των εγγράφων φαίνεται εκ πρώτης όψης επαρκής για να εξασφαλιστεί ένα σαφές, συγκεκριμένο και επαρκές πλαίσιο διαχείρισης. Παρόλα αυτά, η διαχείριση του ισχύου του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας ε, ανέδειξε μια σειρά προβλημάτων που δυσχεραίνουν την ε, σωστή πορεία της ε, λειτουργικότητας των προγραμμάτων. Αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε ως εξής. Καταρχήν, η αοριστία σε ό,τι αφορά τη σημασία και την εμβέλεια πολλών μέτρων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε μάλιστα από την ελάχιστη χρησιμότητα που είχαν τόσο ο εφαρμοστικός κανονισμός όσο και το βατεμέκον που εκατέρτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι δεν υπερβολεί υπερβολή να λέμε ότι και τα δύο έγγραφα δεν ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα για την υλοποίηση των στόχων ε, για τα οποία ε, σχεδιάστηκαν. Ο εφαρμοστικό κανονισμό θα έπρεπε να συμπληρώσει κανονικά ε, τον βασικό κανονισμό, αναλύοντα ε, κάποιε έννοιε ώστε να αποφευθούν ε, αποκλίνουσε ερμηνείε από τι αρχέ που προβλέπει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελίας. Από την άλλη πλευρά, το Βαντεμέκουμ θα έπρεπε να ερμηνεύσει σωστά κάποια άκρα του κανονισμού, για τα οποία ίσω δημιουργούνταν αφιβολίε για την εμβελιά του. Διαπιστώσαμε ότι αυτή η οριστία κατέστη, ε, κατέστη επιτακτική την ανάγκη μιας πληθώρας ερμηνευτικών σημείων ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δημιούργησαν μια τεράστια ανασφάλεια στους ε, διάφορους τομείς που ασχολούνταν με τη διαχείριση των ταμείων. Και μάλιστα το 2011 χρειάστηκε να εκδώσει πολλά τέτοια ερμηνευτικά σημειώματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αρχή διαχείρισης συγκέντρωσε μέχρι και 86 ερμηνευτικά τέτοια σημειώματα και από αυτά 30 εκδόθηκαν γενικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα 56 τέτοια ερμηνευτικά σημειώματα ήταν ερωτήσεις που έθεσε η Ισπανία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι λογικό για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2007 να απαιτούνται τόσε πολλέ εξηγήσει και ερμηνείε όταν έχουν περάσει ήδη δύο τρίτα από την θέση σε ισχύ του. Επιπλέον, η υπερβολική προθεσμία, η μακρά προθεσμία που ε, χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει απαντήσει στα ερμηνευτικά ερωτήματα που έθεσαν τα κράτη-μέλη. Σε μερικέ περιπτώσει άργησε και ένα εξάμεινο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει απάντηση στι ερωτήσει μα και τι απορίε μα. Μερικέ φορέ ε, δεν ε, έχουμε λάβει ακόμη, δεν, έχουμε, δεν λάβαμε καν απάντηση. Περιμένουμε απάντηση σε 13 ακόμη ερωτήσει. Σε ό,τι αφορά τον άξονα 4, τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλληλευτικών ζωνών. Επίσης, ε, είχαμε κάποιες ερωτήσεις ε, για το εμπόριο ε, κάποιων προϊόντων που άμεσα ή έμεσα σχετίζονται με την αλία, την παραγωγή και εμπορευματοποίηση κάποιων ψαριών ενιδρίου, η αγορά από δεύτερο χέρι, η στιοφόρα και ούτω καθεξής. Βλέπετε ότι μπροστά στι θέσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε πολλέ αμφιβολίε για τη χρηματοδότηση και τέτοιων δραστηριοτήτων. Έτσι, περιορίζονται οι δυνατότητε διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των αλλιέων. Και υπάρχει μια αποκαρδίωση, αποθάρρυνση από του διαχειριστέ των μέτρων, που είναι κάποιε τοπικέ ομάδε αλλιέ που βλέπουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν τι πρωτοβουλίε του. Αυτή η καθυστέρηση επίση εμπόδισε τη λήψη αποφάσεων για δράσεις που απαιτούσαν μια άμεση απάντηση εκ μέρου τη διοίκησης. Ένα τρίτο στοιχείο που σχετίζεται άμεσα με τα δύο προηγούμενα αφορά τι ερμηνείε που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ερμηνείε αυτέ ήταν συστηματικά συσταλτικέ ε, σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφάρμοσε την αρχή της καταγράμμα ε, εφαρμογής του κανόνα χωρίς να λάβει υπόψη την έμεση βούληση του νομοθέτη που περιλαμβάνεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένα παράδειγμα από, την, από τον αντίκτυπο που είχε στην ανανέωση του παραγωγικού ιστού αφορά την αγορά ακινήτων που ήδη είχαν κατασκευαστεί και κυρίως αγορά βιομηχανικών σκαφών για την εγκατάσταση κάποιων βιομηχανιών μεταποίησης. Και μάλιστα διαπιστώσαμε ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες ήταν επιλέξιμες για επιχειρήσεις, αρκεί ε, να μην ε, περιλαμβάνονταν νέα μετατόπιση αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν περιλαμβάνονται όμω τέτοια κριτήρια στον κανονισμό. Επιπλέον, τα κριτήρια επιλογή ε, που ενέκρινε η Επιτροπή ε, Παρακολούθηση και είναι γνωστά προβλέπει ότι δεν θα επιχορηγούνται για, το, για την αξία του οικοπαίδου τοπικών αγορών, μια και η αγορά τέτοιων βιομηχανικών σκαφών είναι μια επιχορηγήσιμη χρηματοδοτούμενη δράση. Επίσης, σε μια τέτοια συσταλτική ερμηνεία για τις με δαπάνε σε παραγωγικές επενδύσεις, ε, θα έπρεπε να είναι πιο σαφής η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η απάντηση της Ισπανία, ε, σε ό,τι αφορά την Ισπανία για τα κριτήρια επιλογή, ε, θα έπρεπε να, είναι, να μην δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν ελάχιστη χρήση και της της ε, Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Δεν έγινε επαρκής διαβούλευση με τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, αυτό οφειλόταν στην αοριστία του κανονισμού και στην έλλειψη βούλης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περαιτέρω διαβούλευση με τα κράτη-μέλη. Σε τελική ανάλυση, η Επιτροπή, η Επιτροπή του ΕΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα έπρεπε να είχε πρωταγωνιστικό χαρακτήρα στη διαχείριση ε, του ΕΤΑ έγινε απλώς ένας οργανισμός που συγκέντρωνε πληροφορίες. Ε, κρίμα, γιατί θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να διαμορφωθεί μια κοινή θέση. Ένα πέμπτο στοιχείο που επηρέασε την λειτουργία του ΦΕΠ είναι η απέτηση κομισιών να εφαρμοστούν αναδρομικά ορισμένα κριτήρια που η, η εμβέλειά του ήταν σε για τα κράτη-μέλη. Έτσι δημιουργήθηκε μια τεράστια νομική έλλειψη ασφάλειας, ασφάλεια δικαίου για τα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση κάποιων δράσεων για συγκεκριμένο τομέα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αφισβητήσει συστηματικά τα κριτήρια και τις δραστηριότητες των κρατών μελών. Δεν είναι σαφές. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την συμβολή των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσαρμογή της ικανότητας των αλληλευτικών στόλων στις ισχύουσες αλληλευτικές δυνατότητες. Γιατί είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα. Η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύθηκε το 2011 έχει ως στόχο την ανάλυση του κατά πόσο το ισχύον πλαίσιο για τη μείωση της ελληνική ικανότητας ήταν αρκετά σαφές και αν τα ειδικά μέτρα που υπήρχαν εφαρμόζονταν με το, με, με, ε, δέοντα τρόπο, με αρκετά συγκεκριμένο και απτό τρόπο. Φάνηκε εδώ ένα σοβαρότατο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την, ε, τον ορισμό ενός ε, σημαντικού όρου ε, που ερμηνευόταν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις μεταφράσεις. Για παράδειγμα, στα Ισπανικά αναφερόταν ότι οι επενδύσεις ε, δεν θα έπρεπε να αυξάνουν την ε, αλλιευτική ικανότητα, ενώ στα Αγγλικά αναφερόταν η αλληλευτική the ability of the vessels to catch fish, την ικανότητα των σκαφών να αλλιεύσουν. Επίσης, δεν φάνηκε αν θα έπρεπε να αναθεωρηθούν τα προγράμματα για τις επενδύσεις στα σκάφη, ώστε να αποφευχθούν επενδύσεις που θα δημιουργούσαν αύξηση της ελευτικής δυνατότητας. Επίσης, τι είδου επενδύσεις είναι επιλέξιμες για δημόσιες επιχορηγήσεις. Υπήρχε ασάφεια προς την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Δεκέμβριο του 2011 ε, δόθηκαν γραπτώς κάποιες εξηγήσεις στα κράτη-μέλη επαφίοντας τη δυνατότητα να, ε, να κρίνουν ποιες είναι οι επιλέξιμες ε, επενδύσεις. Για πρώτη φορά αναφέρεται η αρχή ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβαίνουν σε περιπτωσιολογικό προηγούμενο έλεγχο για να κρίνουν κατά πόσο ένας εξυγχρονισμός μπορεί να οδηγήσει αύξηση της ελευτικής ικανότητας. Οπότε περιλαμβάνονται, ε, περιορίζονται κάποιες επενδύσεις και αποκλείονται άλλες ε, που κανονικά θα μπορούσαν να επιτρέπονται. Αυτό δείχνει ακριβώς την αοριστία, την έλλειψη ε, συγκεκριμένου χαρακτήρα του κανονισμού του ΕΤΑ και την έλλειψη λειτουργικότητας κάποιων δομών συντονισμού, όπως είναι η Επιτροπή του ΕΤΑ. Είχαμε λοιπόν μία αναποτελεσματική διαχείριση με κατασπατάληση ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων. Επίσης, στο τελευταίο σημείο τη παρέμβασης θα ήθελα να αναφερθώ στον αντίκτυπο που είχαν οι επανειλημμένοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις ε, στις ε, αρχές διαχείρισης των ταμείων σε αυτή την περίοδο προγραμματισμού. Η αρχή ελέγχου πραγματοποίησε 136 ελέγχους ε, σε σχέδια της ε, Γενικής Διοίκησης ε, του κράτους, ενώ οι ενδιάμεση οργανισμοί επιθεώρησης πραγματοποίησαν 619 ελέγχους στην τοπική αυτοδιοίκηση, για τοπικά σχέδια δηλαδή. 755 έλεγχοι συνολικά έγιναν στην περίοδο 2009-2011. Οι έλεγχοι αυτοί δεν ήταν οι μοναδικοί. 27 επιπλέον έλεγχοι έγιναν για τα συστήματα διαχείρισης. Ε, μια τέτοια πληθώρα ελέγχων όντως ε, εξασφαλίζει μια καλύτερη εκτέλεση ή μήπω αντίθετα από έναν αριθμό και μετά οι συμπληρωματικοί έλεγχοι δεν βελτιώνουν τη διαχείριση αλλά απλώ ε, επιτείνουν την κατασπατάληση οικονομικών πόρων. Νομίζω ότι το θέμα τη ε, διαχείριση και της αποτελεσματικότητας ελέγχου είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη. Για όλου όσου ασχολήθηκαν με τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλία, η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη, διάφορες διοικήσει και οι αποδέκτε των ταμείων και των κονδυλίων αυτών έκριναν ότι το νέο ταμείο θα πρέπει να είναι πιο εύχριστο στην πράξη για να εξασφαλίσει την απαραίτητη συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των βιολογικών ε, και ελευτικών πόρων προκειμένου να καλυφθεί όλη η αλυσίδα και να εξασφαλιστεί μια, ένας βιώσιμος κλάδος αλίας και μεταποίησης. Νομίζω ότι από τα διδάγματα που αντλήσαμε από τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας θα μπορέσουμε να προβλέψουμε ένα πιο ορθολογικό σύστημα για μια πιο εύχρηστη και γρήγορη μελλοντική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλίας. Σας ευχαριστώ. Τραστόη να δώσω το λόγο στην κυρία Κούκα, υπεύθυνη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας στο Φιλανδικό Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομείας. Ο κύριος Κούκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής. Θέλουμε να δούμε τις διαδικασίες της ε, μεταρρυθμιζόμενης αλληλευτικής πολιτικής. Στο κοινοβούλιο μας στη Φιλανδία τα συζητήσαμε αυτά με την αρμόδια Επιτροπή γιατί νομίζω είναι σημαντικό να δούμε και τις δικές μας εμπειρίες και τις γνώσεις που έχουμε αποκομίσει ως σήμερα. Το βασικό μου μήνυμα αφορά το πρότυπο διαχείρισης που προτείνεται για το μελλοντικό ταμείο. Το σημείο αφετηρίας εδώ είναι ότι το Ταμείο Αλίας σήμερα είναι σχετικά μικρό σε όγκο σε σχέση με άλλα ταμεία. Ήταν ευέλικτη η διαχείριση στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και κατάλληλη για ένα τέτοιο είδους ταμείο. Έτσι, έχουμε καλά αποτελέσματα και στον ευρωπαϊκό τομέα. Και ο λόγος ήταν ότι μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε έτσι τις δραστηριότητες και τους πόρους του τομέα, χωρίς να, διασπά... να διασπείρεται ο έλεγχος. Problem εδώ οι πόροι για τους σκοπούς ελέγχου πρέπει να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Το ίδιο και οι ανάγκες του βιομηχανικού τομέα. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι ότι το σημερινό μοντέλο διαχείρισης είναι για μας κατάλληλο. Να προσθέσω βέβαια ότι οι απαιτήσει στο μέλλον προβλέπεται να είναι αυστηρότερες. Αυτό θα έλεγα ότι θα δυσκολέψει τα πράγματα στο μέλλον και από την πλευρά της Επιτροπής και θα συμφωνήσω εδώ απολύτως με τον Ισπανό συνάδελφο. Εδώ λοιπόν χρειάζεται χρησιμότερος τρόπος εργασίας από ότι περισσότερη ποσότητα για, το, για τον τομέα Επίσης, ε, μεγαλύτερη προσπάθεια από τα κράτη-μέλη που έχουν ε, μεγαλύτερων διαστάσεων προγράμματα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κοινέ διατάξεις για το Ταμείο προβλέπει να αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης ε, κατά τρόπο που να προσωμιάζει αυτό της, το Ταμείου Περιφερει... της Ανάπτυξης της Υπέθρου. Θα πρέπει όμως να δούμε αν είναι κατάλληλοι οι κανόνες αυτοί διαχείρισης, διότι εκείνο το ταμείο, όπως και το κοινωνικό ταμείο και το ταμείο συνοχής, μπορούν να διατηρήσουν τα υπάρχοντα μοντέλα τους. Δεν υπάρχει λόγος προσαρμογής και του αλληλευτικού ταμείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει πει ότι θα υπάρξουν σχέσει συνεργασία και εξοικονομήσεις σε διοικητικό επίπεδο εφόσον ακολουθεί το ίδιο μοντέλο από όλα τα ταμεία. Όμω, αυτό το συζητήσαμε με τον ε, φορέα πληρωμών ε, στη Φινλανδία που είναι υπεύθυνο για το Ταμείο Ανάπτυξη τη και είπε ότι θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι και δεν μπορεί να ε, ξέρει που θα γινουν οι εξοικονομησει ακριβω με το νεο συστημα ουτω η αλλω και η διαχειριση του ταμειου αναπτυξη τη επεθρου ειναι καποιε φορε επαχθη λογω των απαιτησεων που θα αυξηθουν και νέων αρμοδιοτήτων που θα ανατεθούν στο προσωπικό του. Επίση, η εμπειρία μα ω τώρα δείχνει ότι οι πληρωμέ προ του αλληλεί και άλλου δικαιούχου θα δυσκολέψουν και θα καθυστερούν. Σήμερα, οι πληρωμέ από το Ταμείο ε, Αλία έρχονται σχετικά σύντομα. Οι Γεωργοί όμω περιμένουν περισσότερο για τι πληρωμέ από το Ταμείο Αναπτύξη τη Πέθρου. Έτσι λοιπόν οι σχέσει συνεργασία σε πρώτη όψεω μπορεί να φαίνονται θετικέ. Όμω τελικώ από τη δική μα την πλευρά φαίνεται να μην είναι εφικτέ μακροπρόθεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι υπάρχουν πετυχεμένα παραδείγματα από τον τρόπο διαχείριση, το μοντέλο διαχείριση του Ταμείου Ανάπτυξη τη Υπέθρου. Εγώ νομίζω όμω ότι το έβριμα αυτό τη Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το μοντέλο αυτό δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Τα κράτη-μέλη που θα θέλουν τέτοιο σύστημα διαχείριση να το προβλέψουν, να το κάνουν εθελούσια, βάσει των ε, ισχυρών των κανόνων. Υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα με τις προτάσει τη Επιτροπής. Ο έλεγχο των επιδόσεων. Τα κονδύλια δηλαδή που θα αποδίδονται στα κράτη-μέλη μόνο να αποτιμηθούν οι επιδόσεις των προγραμματών τους. Αυτό αν το δούμε στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού θα δούμε ότι δεν ήταν τόσο καλή η ιδέα. Ήταν μια παχθής διαδικασία, χωρίς ιδιαίτερη προστιθεμένη αξία. Τώρα γιατί να δουλέψει αυτή τη φορά. Ουσιαστικά θα αυξηθεί το διοικητικό άχθος. Και βεβαίως ο διοικητικός φόρτος για τα κράτη-μέλη. Εδώ να πω λίγα λόγια για την ουσία της πρότασης περί Ταμείου Θάλασσας και Λίας. Νομίζουμε η υδατοκαλλιέργεια είναι ένα γοργά αναπτυσσόμενο τομέα στα πλαίσια τη Αλλίας. Επιτρέπει την παραγωγή περισσότερων ψαριών σε μεγάλε ποσότητε. Και μάλιστα σε περιοχέ που τα αποθέματα μπορεί να είναι σπανιότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω δεν έχει σημειώσει ότι το μέσο αυτό δεν αναπτύχθηκε εξίσου γοργά στην Ευρώπη που σε άλλα μέρη του κόσμου. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το καλό του τομέα αυτού, διότι λείπουν η κάλυψη των αναγκών, ε, λείπει η κάλυψη των αναγκών στη νέα πρόταση. Λόγω χάρη επενδύσεις σε αλία που δεν θα είναι παράκτεια. όπως το παράδειγμα της Φινλανδίας που σεβόμαστε και τους περιβαλλοντικούς κανόνες με συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για την, υδατοκαλλιέργεια. Και αλλα κάτι κράτη-μέλη έχουν εντοπίσει τις δικές τους ανάγκες για την υδατοκαλλιέργεια που όμως λείπουν και δεν καλύπτονται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά δεύτερον, θα πρέπει τα πορίσματά μας για την υδατοκαλλιέργεια να τα εφαρμόσουμε προκειμένου να, εφαρμόσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε για έρευνε που να επιτρέψουν την ανάπτυξη του τομέα. 18 κράτη-μέλη έχουν υποβάλει κοινή πρόταση, η οποία θέλαμε να ληφθεί υπόψη από την τοποθέτηση του Συμβουλίου. Τα κράτη-μέλη λοιπόν με την Προεδρία του Συμβουλίου βλέπουν κατά πόσο δικέ προτάσει είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή για την προστασία του τομέα αυτού στην Ευρώπη επίσης. Με την εικόνα αυτή να θυμίσω ότι η σύγχρονη υδατοκαλλιέργεια είναι πραγματικά υψηλή τεχνολογία κλάδο. Οι δραστηριότητε οι περισσότερε είναι αυτοματοποιημένε και σε τέτοιε περιοχέ, μονάδε παραγωγή, μπορούμε να συνδυάσουμε την υδατοκαλλιέργεια με ε, γεωργία θερμοκηπίου καλλιέργεια θερμοκηπίων και με χρήση πράσινων μεθόδων, οικολογικών μεθόδων. Μειώνεται έτσι και ο όγκος των ε, απορριμμάτων και αποβλήτων και νομίζω ότι τέτοιου είδους ε, επενδύσεις και πρωτοβουλίες πρέπει να τις στηρίξουμε και στο μέλλον. Αλία. Η αλία ήταν βεβαίως πάντοτε στο επίκεντρο των αλληλευτικών δραστηριοτήτων όμως ε, ε, το μέσο αυτό έχει γίνει τόσο αποδοτικός που απειλούνται τα αλληλευτικά αποθέματα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και αλλού. Εάν δει κανεί ε, τα πολιτικά συμπεράσματα που θα πρέπει να αντλήσουμε, θα φανεί ότι οι ανάγκε κάθε κράτου μέλου διαφέρουν μεταξύ του. Στην Βαλτική θάλασσα, λόγω χάρη για τη Φινλανδία, τα αλληλευτικά αποθέματα βρίσκονται σε σε καλή κατάσταση και θα μπορούσε να μειωθεί και το κόστο τη αλεία χωρί να κινδυνεύσουν τα αποθέματα. Στην Φιλανδία, επίση στα εσωτερικά ύδατα με 100.000 λίμνε, έχουμε εκατοντάδε είδη ψαριών που μπορούμε να αλλιεύσουμε και εκεί. Η αλεία λοιπόν αυτή ε, των ιστορικών υδάτων είναι εξίσου σημαντική με την θαλάσσια. Υπάρχουν βεβαίω διαφορετικά προβλήματα με τα αλλιευτικά αποθέματα από χώρα σε χώρα. Στη Φινλανδία είχαμε μεγάλο πρόβλημα με τις φώκες οι οποίες κατέστρεφαν τα δίχτυα και βεβαίως χάνονταν έτσι πολλά αλλιεύματα. Είναι σημαντικό για τους Φινλανδούς αλλιείς να στηριχθούν με κονδύλια και να κάνουν επενδύσεις ώστε τα παραδοσιακά τους ε, εργαλεία να βελτιωθούν και να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς κρατική βοήθεια. Επίση. πρέπει να στηριχθούν και οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα αυτό. Λίγοι είναι οι νέοι που είναι τόσο τολμηροί, ώστε να ξεκινήσουν μια καριέρα ως αλληλείς. Τέλος, να σας δείξω κάποιες εικόνες που απεικονίζουν τις ειδικότερε συνθήκες της Φινλανδίας στον τομέα της αλίας. Εδώ βλέπετε μια εικόνα της λίμνης Αριτουρμάγκη, σημαντική για τους Φινλανδούς αλλοίες ή την αλία στο, το χειμώνα, στους πάγους. Που αυτό για μας μπορεί να γίνει και στη θάλασσα και σε νερά λίμνης. Είναι σημαντικό εδώ να εξοπλίσουμε τους Φινλανδούς με, τον απαραίτητο, με τα απαραίτητα εργαλεία και για τη θαλασσιαλία και για την αλία στις λίμνες. Και φυσικά αυτή η χειμερινή αλία έχει και μεγαλύτερο κόστος για του αλίες και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τέλος, βλέπετε πόσοι οι γκρίζε φώκες μπορούν να γίνουν ε, αρπακτικά, απειλητικά αρπακτικά που ε, θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την αλία. Ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί πολύ την τελευταία δεκαετία και αυτό είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο για τους Φινλανδούς ε, ψαράδες, αλλά και για λύσεις στις υπόλοιπες χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κούκα. Για τις φώκες έχουμε ακούσει πολλά και από τον κύριο Χάγκλαντ. Τώρα, να δώσω το λόγο στην κυρία Σφετάνκα Γιαντζέβα Παλάσοβα, <coughs> διευθύντρια του Διευθυντηρίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας και της, ε, Εθνικό Φορέα για την Αλία και τις Αυτοκαλλιέργειες. ΝΑΦΑ. Dear Mr. Chairman. Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να συμμετάχω εδώ σε αυτή την Επιτροπή και να σας παρουσιάσω την εμπειρία μας στις δυσκολίε διαχείριση του προγράμματος και να σας παρουσιάσω τις προτάσεις της Βουλγαρίας για το νέο κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλίας. Η Εθνική Υπηρεσία Αλίας και Ιδατοκαλλιέργειας είναι η αρμόδια αρχή που χειρίζεται αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ζωτική σημασία για τη χώρα μας. Μετά, ε, από τη στιγμή που η Βουλγαρία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπειρία μας λοιπόν στη διαχείριση είναι αυτή που θα σας παρουσιάσω. Πρωτού όμως αρχίσω, θα ήθελα να κάνω μια περίληψη της ισχύουσα κατάστασης στον τομέα της αλληλεία. Στην Βουλγαρία έχουμε 230 2.336 αλληλευτικά σκάφη, 339 φάρμες υδατοκαλλιέργεια και 37 επιχειρήσεις επεξεργασίας ε, προϊόντων αλληλεία και υδατοκαλλιέργεια. Αυτά είναι τα δεδομένα του αλληλευτικού μαστόλου στόλου και τα δεδομένα για τι ε, φάρμες υδατοκαλλιέργεια. και ορισμένα δεδομένα για τις ε, επιχειρήσεις επεξεργασίας αλλιευμάτων. Εντοπίσαμε προβλήματα στο μέτρο 1-1 στην ε, δημόσια βοήθεια για την μόνιμη πάυση των αλληλευτικών δραστηριοτήτων και επίσης εντοπίσαμε ότι προσοχή δίδεται στο μέτρο 2.1 τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και το μέτρο 2.6 τις επενδύσεις στην επεξεργασία και το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων αλίας και των ε, προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Μέχρι τώρα οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί είναι 103 και η αξία τους ανάρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ βρίσκεται σε διαδικασία έγκριση, βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης 38 συμβάσεις με αξία 6,2 εκατομμυρίων ευρώ. Δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά για τις πλήρωμες που είναι περίπου το 14%, 14 εκατομμύρια ευρώ Και για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό, οι αρμόδιες αρχές στοχεύουν να προωθήσουν μέτρα για την πληροφόρηση του κοινού. Επίσης, συνεργαζόμαστε στενά με τους αντιπροσώπους όλων των ενδιαφερομένων στον τομέα αυτό, αλλά και με άλλα διοικητικά σώματα στη χώρα και με τους επενδυτές. δυσκολίες τώρα που έχουν αντιμετωπίσει οι αρμόδιες αρχές. πρώτη ομάδα είναι οι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή του προγράμματος. Η έναρξη του προγράμματος συνέπεσε με την έναρξη της οικονομικής κρίσης και κατέστησε δύσκολη την πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Η χρηματοδότηση λοιπόν έπεσε κατά 50% και αυτό δυσκόλεψε πολύ τις επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αυξήθηκε η παραοικονομία και υπήρξε σημαντική δυσκολία στον έλεγχο των ε, δραστηριοτήτων της παραοικονομίας. Τέλος, ο παράγοντας επίσης που επηρέασε την εφαρμογή ήταν η ανεργία, τα επίπεδα ανεργίας, το κόστος των καυσίμων και η ζήτηση, η μειωμένη ζήτηση προϊόντων αλίας. Επιπλέον, ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες ε, που δραστηριοποιούνται στην, Ευρωπαϊκή, στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δυσχέρανε περισσότερο τα πράγματα. Στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία η κατάσταση στον ε, τομέα της αλίας είναι παρόμοια και θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε και τις απόψεις των άλλων κρατών μελών για, την, για, τον, για τις δικές και τις δικές τους εμπειρίες. Μετά, ένα άλλο πρόβλημα για την Βουλγαρία είναι οι κανόνες και, ο σαφής, και η έλλειψη σαφούς ορισμού κανόνων και ρυθμιστικών μέτρων. Οι επόμενοι παράγοντες έχουν να κάνουν με το έργο των, ε, αρχών, των αρμόδιων αρχών. Εμείς κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής δεν λάβαμε χρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό όργανο. Και επιπλέον δημιουργήθηκε και αρκετός διοικητικός φόρτος που δυσχέρανε το έργο μας. Επίσης, η καθυστερημένη έναρξη του προγράμματος στη Βουλγαρία οδήγησε στη μείωση των διαθέσιμων κονδυλίων. For bigger investment projects. Επίσης θα επανεξετάσουμε όλα τα project που τρέχουν και, θα, και επιθυμούμε να αυξήσουμε το ποσοστό των ε, προκαταβολικών πληρωμών. Όσον αφορά την, ε, τον έλεγχο, εντοπίσαμε ορισμένους, ορισμένα προβλήματα δυσκολίες από την πλευρά των δικαιούχων τώρα υπήρξαν δυσκολίες στην παροχή χρηματοδοτικών μέσων για την εφαρμογή των προτάσεων αυτών των project. Μετά ε, υπήρξαν το καθεστώς, το διοικητικό και το ρυθμιστικό καθεστώς ήταν αρκετά περίπλοκο όσον αφορά τον έλεγχο και τις ε, απαιτήσει για την υγιεινή και επίσης ο διοικητικός φόρτος ήταν και εδώ αρκετά μεγάλος. όσον αφορά τις προτάσεις για την βελτίωση του κανονισμού για το νέο Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, η Βουλγαρία έχει την ακόλουθη θέση. Υπάρχει, πιστεύουμε, ανάγκη για κατασκευή νέων λιμένων ε, τόπων εκφόρτωσης με βοήθεια χρηματική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ο νέος κανονισμός χρειάζεται σαφείς ορισμούς και σαφή ρύθμιση της εφαρμογής τους, ενίσχυση των μέτρων συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης καλωσορίζουμε την, ε, την προσπάθεια για προώθηση νέων μορφών ε, υδατοκαλλιέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας αυτής. Πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα όχι μόνο στις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας που θα γίνουν, αλλά και σε αυτές που ήδη λειτουργούν. Η υδατοκαλλιέργεια είναι πολύ σημαντική για τη Βουλγαρία και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτή τη χώρα μέσα στην, ε, κατά τη νέα ε, περίοδο προγραμματισμού. Πιστεύουμε ότι το 50% είναι πολύ χαμηλό ποσοστό για την χρηματοδότηση, τη μέγιστη χρηματοδότηση και θα έπρεπε να αυξηθεί στο 60%. Προτείνουμε να συμπεριληφθεί μια διάταξη για επιμήκυνση της περίοδου αυτόματης αποδέσμευσης και την εφαρμογή ενός επαρκούς μηχανισμού για, την, ε, για τον έλεγχο της, ε, ενός λογιστικού κώδικα και του συστήματος των δικαιούχων. Συμπεραίνοντας λοιπόν, Ελπίζουμε να λάβετε υπόψη ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι νέα κρατημέλη και ω νέα κρατημέλη δεν είχαν τον, το ίδιο χρονικό περιθώριο για να αποκτήσουν εμπειρία και να επιτύχουν αυτά αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι οι προτάσεις μας για τον νέο κανονισμό θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ελπίζουμε ότι στη νέα προγραμματική περίοδο η Βουλγαρία θα επιτύχει περισσότερη ανταγωνιστικότητα και περισσότερη βιωσιμότητα στον τομέα της Ελίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και ευχαριστώ τους τρεις πρώτους ομιλητές σήμερα το πρωί. Έχουμε προπλέψει χρόνο για συζήτηση βάσει των τριών αυτών παρουσιάσεων και θα ήθελα να καλέσω τα μέλη της Επιτροπής που θέλουν να παρέμβουν να μας το πούν. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι τρεις πρώτοι μιλητές για σήμερα το πρωί επανέλαβαν ότι το σημερινό σύστημα είναι πολύ περίπλοκο ούτως ή άλλως. Είναι δυσνόητοι κανόνες για τις επιλέξιμες πληρωμές και καθυστερούν πολύ οι διευκρινήσεις από την πλευρά της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν στη συνέχεια, μάλλον και η Επιτροπή να το σχολιάσει αυτό, αλλά κατά πρώτα να δώσω το λόγο στην κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες ε, οι ομιλίες των τριών εμπειρογνωμόνων που μίλησαν για τις αδυναμίες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας και την ε, συνέχιση, από ό,τι φαίνεται, των προβλημάτων ε, με τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μελλοντικό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει εξηγήσει και να απαντήσει σε όλες αυτές τις επικρίσεις που ακούσαμε έλλειψη ελαστικότητας, φοβερή κολλησιεργία σε ό,τι αφορά την έκδοση των ερμηνευτικών σημειωμάτων. Όπως είπε ο εκπρόσωπος της Ισπανίας, πολλές φορές εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης εμποδίστηκαν προγράμματα του άξονα 4, της διαφοροποίησης και ούτω καθεξής. Επίσης, ε, είναι άνω ποταμών η εφαρμογή της αναδρομικότητας. Η αναδρομικότητα είναι η έσχατη λύση ε, στο δίκαιο. Και έχουμε νομικούς που μπορούν να μας το εξηγήσουν. Αν είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χρησιμοποιεί την αναδρομικότητα πολύ πιο συχνά από ό,τι είναι απολύτω απαραίτητο, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Επίση, αναφέρθηκε η έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων, η αοριστία ω προ τα μέτρα. Από την άποψη αυτή, ο κανονισμό είναι διπλά περίπλοκο, γιατί είναι διπλή αοριστία. Πρώτον, λείπουν κάποια μέτρα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν, αλλά και η αοριστία είναι σημαντική αδυναμία. Αν στο παρελθόν είχαμε προβλήματα με την αοριστία, είναι ακόμη σημαντικότερο το πρόβλημα με τον τρέχοντα κανονισμό. Ιδιαίτερα το, η παράγραφος για τι οργανώσει παραγωγών. Δεν ξέρουμε τι θα χρηματοδοτηθούν, ποιε είναι οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράση και ποιε όχι. Φαίνεται ότι οι οργανώσει παραγωγών θα πρέπει να διαχειριστούν και το ζήτημα των απορρίψεων. Έχουν πολύ περισσότερε αρμοδιότητε δεν φαίνεται με σαφήνεια από την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι επιδέχεται χρηματοδότηση και τι όχι. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μην περάσει απαρατήρητο, να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλες αυτές τις ε, κριτικές και να μας πει αν με τη νέα πρόταση βελτιώνεται η κατάσταση. Γιατί έχω την αίσθηση ότι με τη νέα πρόταση αντί να βελτιωθεί επιδεινώνεται η ισχύουσα κατάσταση. Ευχαριστώ κύριο Σκούν. Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Φράγκε αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πράγματα και θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορούμε να έχουμε κάποια απάντηση πάνω σε αυτά, γιατί η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη. Έχουμε πολλά ερωτήματα. Πώς θα, πώς θα διαχειριστούμε το Ταμείο, πώς θα διαχειριστούμε διοικητικά. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω μια απάντηση. Γίνεται αυτό. I think maybe... Νομίζω ότι το να δώσουμε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, όχι μόνο αυτά που τέθηκαν από τους ομιλητές πριν, αλλά και από τα μέλη της Επιτροπής. Πρέπει να ακούσουμε όλα, όλες τις ερωτήσεις πρώτα. Κύριε Κούν, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ναι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω για τους τρεις ομιλητές από την Ισπανία, τη Φιλανδία και τη Βουλγαρία. Πραγματικά ήταν εκτενείς παρουσιάσεις. Υπήρξαν ορισμένα σημεία τα οποία θέλω να θίξω έχουν ζωτική σημασία για το Ταμείο και το μέλλον του Ταμείου τα επόμενα 7 χρόνια. Από την πλευρά της Ισπανίας αναφέρθηκε ρητά ότι εάν η Κομισιόν θέλει να δώσει κάποια ε, χρηματοδοτικά μέσα, πρέπει να γίνει μείωση του αλληλευτικού στόλου. Πιστεύω πως είναι αναγκαίο επιτέλους να έχουμε πληροφορίες από την Eurostat ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία για το μέγεθος του αλληλευτικού στόλου, για την ε, αλληλευτική δυνατότητα του αλληλευτικού ε, μας στόλου, στα επιμέρους κράτη-μέλη να έχουμε λεπτομερή στοιχεία και μετά θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αυτά που μας είπε ο συνάδελφος Αλάν Καντέ και να δούμε τι δυνατότητες θα έχουμε στο μέλλον με, με σύγχρονα μηχανήματα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ποσοστώσεις, να μπορέσουμε να επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, να δώσουμε βάση στην περιβαλλοντική και οικολογική διάσταση είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Είναι κεντρικό το ζήτημα. Τώρα για την υδατοκαλλιέργεια. Αυτή η πρωτοβουλία θεωρώ πως είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει η αλλιευτική δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη στις ε, θαλάσσιες περιοχές αλλά και στα εσωτερικά ύδατα να, να χρησιμοποιούνται με τον ε, περισσότερο αποδοτικό τρόπο. Και η πρόταση της Επιστροπής για το νέο ταμείο αναφέρεται σε επενδύσεις, αλλά μόνο στον, τομέα, στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν ε, όμως και άλλοι τομείς και η παράκτια ε, και, και, όχι μόνο από, τον, από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα. Χρειάζεται να έχουμε ερεθίσματα, να υπάρξουν έρευνες από ερευνητικά ιδρύματα για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλά και αποδοτικά τη γνώση μας στην Αλία και στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Τώρα επενδύσεις, αυτό που ανέφερε η συνάδελφος από τη Βουλγαρία, υποδομή χρηματοδότηση για την αλληλεία. Μπορούμε να το συνδέσουμε αυτό με τα διαρθρωτικά ταμεία. Και είναι αναγκαίο να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Και να δούμε πώς θα λειτουργήσει στο μέλλον το ταμείο. Επίσης, ο συνάδελφος από την Φιλανδία ανέφερε τους γόνους των ψαριών και πώς θα τους προστατεύσουμε για να συνεχίσουμε να έχουμε αλλιευτικά αποθέματα, αναφέρθηκε σε ποσοστώσεις, σε λογικές ποσοστώσεις, σε λογικές λύσεις. Και αυτό επίσης είναι κάτι που δεν πρέπει να παραβλέψουμε και θα τελειώσω εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ τι, πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε με τον αυξανόμενο αριθμό των, ε, των ε, ε, θαλάσσιων πτηνών και της εφόκιας. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι η φιλανδική πλευρά έκανε εξαιρετικό έργο και συγγνώμη ε, που έτσι επενέβησα τόσο αυθόρμητα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούν. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκρομπάρτσικ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε στις εισαγωγικές σου παρατηρήσεις ο κύριος Αλάν Καντέκ κατά την έναρξη της ε, δημόσιας ακρόασης. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αιλίας, του νέου ταμείου. Έχουμε διαφορετικούς σκοπούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στην ε, προβλέπει από ό,τι φαίνεται στη μείωση για να μην πω στην ε, εξαφάνιση <laughs> μερικές φορές της αλίας. Ενώ δικός μας στόχος είναι η υποστήριξη της αλίας, η ανάπτυξη του αλλιευτικού κλάδου. Και Φάνηκε αυτό και από τις ομιλίες των πυρογνωμόνων και των καλεσμένων μας. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε τον αλληλευτικό κλάδο της αλληλείς και ιδιαίτερα τους νέους αλληλείς, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ των γενναιών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μικρή κλίμακα αλληλείας. Γιατί δεν υπάρχει τέτοια συνέχεια μεταξύ γενναιών, δεν θα επιβιώσει αυτή η μικρή κλίμακος αλληλεία. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να στηρίξουμε την ε, μικρή παραδοσιακή αλία, το να εξυγχρονίσουμε τα ελευτικά σκάφη και να βελτιώσουμε την ασφάλεια. Μερικές φορές ε, διακόπτεται η συνέχεια μεταξύ των γενεών αλλιέων και αυτό επιδρά αρνητικά στον αλιευτικό κλάδο. Γι' αυτό θα πρέπει να θέσουμε την ερώτηση είναι πα, παρόμοιοι οι στόχοι δικοί μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή είναι τελείως αντιφατικοί οι στόχοι σε ό,τι αφορά τη στήριξη των Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του Φιλανδού εκπροσώπου, ήταν πολύ επαναστατικές οι διαπιστώσεις που έκανε για την πολύ καλή κατάσταση των αλλιευτικών αποθεμάτων της Βαλτικής. Είναι κάτι που έρχεται σε αντίφαση με αυτό που ακούμε από τις παρουσιάσεις ή και που φαίνεται στην κοινή γνώμη ότι είναι καταστροφική η κατάσταση των αποθεμάτων στην Βαλτική και ότι θα πρέπει να διαλύσουμε τον αλληλευτικό κλάδο στη Βαλτική, επειδή απειλούνται τα λευτικά αποθέματα. Επίση το θέμα τη φώκια και παρόμοιων θηρευτών. Ε, τέτοιοι θηρευτέ, φώκιε, κορμοράνοι, πραγματικά έχουν ολέθρια επίδραση στην κατάσταση των αλληλευτικών αποθεμάτων. Θα πρέπει να αξιολογηθεί λοιπόν η επιρροή του ε, ε, και όπως είπε και ο κύριο Κούν να δημιουργηθούν κάποια προγράμματα διαχείρισης που θα λαμβάνουν υπόψη και αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα των θηρευτών, αυτών των φυσικών εχθρών των ψαριών. Αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο της Φιλανδίας ε, και το θέμα της υδατοκαλλιέργειας που είναι πολύ διαφορετική σε κλειστέ υδάτινε λεκάνε ε, και άρα θα πρέπει να τύχει διαφορετική μεταχείριση από την παραδοσιακή υδατοκαλλιέργεια σε πιο ανοιχτέ θάλασσε. Να υπάρξει λοιπόν διαφοροποιημένη μεταχείριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε κύριε Κομπάτσο. Ο κύριο Ρωμέβα. Uh, um, Ευχαριστώ πολύ. Ε, το δικό μου πρόβλημα είναι πρόβλημα προτεραιοτήτων και όχι περιεχομένου. Διάβασα την πρόταση της ε, Κομισιόν και καταρχάς με προβληματίζει βαθύτατα το γεγονός ότι καθώς φαίνεται υπάρχει μια μαγική λύση για την αλία και αυτό είναι η υδατοκαλλιέργεια και το επαναλαμβάνουμε σαν μάντρα τελευταία. Το ακούμε ξανά και ξανά και ξανά, λες και αυτό είναι η λύση για την αλία αντί να σκεφτούμε ότι η πραγματική και αληθινή λύση είναι στην βιομηχανία αλληλεία. Είναι θέμα λοιπόν προτεραιοτήτων. Και, αλλά όμω ε, αυτό αποφασίζει πού θα πρέπει να τοποθετηθούν τα κονδύλια. Κατανοώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα για τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, ε, ότι είναι για να γίνει βιώσιμη, για να ε, είναι φιλική προς το περιβάλλον. Όμως, Πραγματικά ανησυχώ, διότι επικεντρώνουμε όλες μας τις προσπάθειες, προσπαθώντας να δικαιολογήσουμε κάτι το οποίο ίσως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Κατανοώ ένα μέρος της συζήτησης, αλλά όχι το γενικό σκεπτικό της. Μετά, κατόπιν των σχολείων που άκουσα, βλέπω ότι υπάρχει, υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή του προγράμματος και αυτό συζητείται. Ε, φυσικά δεν είμαι η Δήμον, οπότε δεν μπορώ να αμφισβητήσω αυτά που μας είπαν οι αρμόδιοι. Όμως, ε, η ερώτησή μου στους τρεις προηγούμενους ομιλητές, δύο προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι η έλλειψη επιστημονικών δεδομένων και μήπως θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούμε στην βελτίωση των επιστημονικών δεδομένων και της επιστημονικής γνώσης και να διοχετεύσουμε τα κονδύλια εκεί. Και αντί να επικεντρωθούμε λοιπόν στους λιμένες, τα σημεία εκφόρτωσης, πιστεύω πως θα πρέπει να δώσουμε βάρος αλλού και έπειτα όσον αφορά την επιστημονική, τις επιστημονικές γνώσεις. Σίγουρα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε στη χάραξη πολιτικής. Τέλος, πιστεύω ότι δεν θύχτηκε πουθενά το θέμα της υπερβάλλουσας αλληλευτικής δυνα... δυνατότητας, της υπεραλίευσης. εάν θέλουμε να βελτιώσουμε το ισχύον σύστημα. Δεν γίνεται να επιχορηγούμε την υπερβάλλουσα αλληλευτική δυνατότητα και αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ. Και σημασία πρέπει να δώσουμε στην μείωση αυτής της αλληλευτικής δυνατότητας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Συμφωνώ και εγώ πως ε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτά που έχει να πει η Επιτροπή. Καταρχάς όμως, θα θέλω να πω ότι έχουμε να κάνουμε με 6.500 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτή την εποχή στην Ευρώπη συζητείται έντονα το πώς θα ξοδέψουμε τα δημόσια χρήματα. Ε, βρισκόμαστε στη μέση μιας οικονομικής κρίσης και πολλοί πιστεύουν ότι τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα και στην καινοτομία και στην ανάπτυξη. Και ότι οι επιχορηγήσεις με την έννοια που είχαν μέχρι τώρα είναι κάτι πεπερασμένο. Δεν βοήθησαν. Δεν βοήθησαν στην ε, γεωργία, δεν βοήθησαν στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Αλλά αν έβγαλε τα ακουστικά και αυτό πάει για σένα, αυτό που λέω. Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι τα δημόσια κονδύλια πρέπει να ξοδεύονται με τρόπο ώστε να βοηθούν το κοινό καλό. Και η πρόταση της ε, Επιτροπής για τα κονδύλια, ότι πρέπει αυτά να δίδονται σε χώρες που συμμορφώνονται με τους κανόνες της κοινή πολιτικής. Είναι θεμελιώδες αυτό, είναι πολύ βασικό. Και σίγουρα υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τώρα ή στο μέλλον που θα διαμαρτυρηθούν ή διαμαρτύρονται ήδη για τους ελέγχους ως προς το που πάνε αυτά τα χρήματα. Όμως, αυτό, αυτή είναι μια απέτηση που προέρχεται από τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν θέλουμε να ξοδεύουμε χρήματα για ε, ε, επιχειρήσεις που είναι βλαβερές προς το περιβάλλον, αλλά τα δημόσια κονδύλια πρέπει να πηγαίνουν μόνο σε δραστηριότητες για το κοινό καλό. Και σε αυτό το σημείο να συμφωνήσω με τον Φιλανδό συνάδελφο πως η υδατοκαλλιέργεια, η φάρμες υδατοκαλλιέργειας είναι κάτι σημαντικό. Έχω δει αρκετά, αρκετές τέτοιες φάρμες στην Σουηδία όπου γίνεται η υδατοκαλλιέργεια αλλά και η επανεξαγωγή ψαριών στο φυσικό τους περιβάλλον. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι ένα άριστο παράδειγμα δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι πραγματικά βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Μετά, πρέπει να αναφερθώ στις φώκες. Ναι, όλοι εδώ σε αυτή την επιτροπή φαίνεται πως ξεχνάνε ότι υπάρχει μια έκθεση. Είχαμε εμπειρογνώμονες από 5-6 διαφορετικές χώρες σε αυτή την επιτροπή οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι οι φώκες δεν επηρεάζουν τα αλληλευτικά αποθέματα στο σύνολό τους. Φυσικά υπάρχουν επιμέρους περιοχές όπου ορισμένες, ε, ομάδες από φώκες ειδικεύονται στο να πιάνουν για παράδειγμα σολομούς. Αλλά έχουμε τεχνολογία για να τις τρομάξουμε, για να τις διώξουμε. Αλλά Όσον αφορά το αν είναι άγριοι θηρευτέ, εγώ μπορώ να σα πω ότι μένω σε περιοχή που έχει φώκε κοντά και ποτέ δεν μου έχει επιτεθεί καμία. Ίσως στη Βαλτική είναι πιο λογικές και συνετές οι φώκε. κυρία... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τους τρεις ομιλητές. Χαίρομαι που ήρθατε εδώ σήμερα διότι έχουμε κάτι καινούργιο. Από τον Δεκέμβρη του 2009 συμμετέχουμε στη διαδικασία συναπόφασης. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, τώρα και το Κοινοβούλιο, έχει δικαίωμα συναπόφασης και νομοθεσίας. Μέχρι πρότινος, η Κομισιόν και το Συμβούλιο μόνο ήταν αρμόδιοι για αυτά τα θέματα και πιστεύω ότι αυτό δίκησε σε αρκετά λάθη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι πολύ καλό που έχουμε αυτή την δυνατότητα. Τώρα, επιμέρους ε, ζητήματα. Είπατε ότι νομίζετε πως η Κομισιόν δεν συμβουλεύτηκε αρκετά τα κρατημέλη και την Επιτροπή, την Επιτροπή εδώ. Ε, δεν ξέρω για την Κομισιόν, αλλά η Επιτροπή εδώ εργάζεται διαρκώς και πολύ σκληρά και πολύ στενά με τα κράτη-μέλη. Έχουμε πάντα εμπειρογνώμονες, καλούμε από το Συμβούλιο, από τα κράτη-μέλη, οι οποίοι μας ενημερώνουν, μας συμβουλεύουν έτσι ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όσον αφορά την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, κατέστησε σαφές ότι οι επιχορηγήσεις δεν πρέπει να δίδονται για την αγορά νέων πλοίων. Στο παρελθόν έγινε αυτό. Έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη αυτή η επιχορήγηση, η οποία σκόπευε στην μείωση του αλληλευτικού στόλου και όχι στην ανανέωση. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε πλέον αυτόν τον ορισμό, διότι δεν αναφέρεται στον ίδιο στόχο. Μετά, είναι σημαντικός ο βέλτιστος έλεγχος. Δεν, δεν υπάρχει υπερβολικός έλεγχος. Αναφέρατε 950 περιπτώσεις ελέγχου, όμως πρέπει να δούμε ποια συστήματα ελέγχου πραγματικά εφαρμόζονται στην ουσία. Ξέρω για παράδειγμα ότι στον τομέα της γεωργίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ελέγξει αυτούς, αυτές τις μεθόδους και τριπλασιάστηκαν στα επιμέρους κράτη-μέλη. Σε εμά στη Γερμανία με το ποσπονδιακό σύστημα έχουμε πολλές επιτρο... επιτροπές και κάθε επιτροπή επιμέρου κρατήδιο ελέγχεται από μια ανώτερη επιτροπή. χρειάζεται να είναι ο έλεγχο, ο ευρωπαϊκός έλεγχος διαφανής, ξεκάθαρος και εξονυχιστικός. Έπειτα, ο κανονισμός πρέπει να συνταχθεί έτσι ώστε να είναι άμεσα εφαρμόσιμος. Κύριε Κούκα από τη Φιλανδία τώρα, είπατε ότι θα είναι δύσκολο να συνδυάσουμε όλα τα ταμεία, το Ταμείο Λίγια, τα διαρθρωτικά ταμεία. Θα υπάρξουν δυσκολίες στην εφαρμογή και στην χρήση και στο συνδυασμό τους. Όμως το παρελθόν δεν ήταν καν δυνατόν να συνδέσουμε αυτά τα ταμεία. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε καν. Ήταν δύσκολο να δούμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ενός, του άλλου. Υπάρχουν αρκετές ε, επικαλύψεις. Πιστεύω λοιπόν πως πρέπει να εξετάσουμε τα αρμόδια ταμεία λεπτομερώς και να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε επικαλύψεις και να τα χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Και πώς μπορούμε να τα οργανώσουμε καλύτερα. Και είναι καλή ιδέα, λοιπόν, να εξετάσουμε τα ταμεία στο σύνολό τους. Χρειαζόμαστε μετά περισσότερη έρευνα, σαφώς. Το λέγαμε ανέκαθεν αυτό. Θέλαμε να συμπεριλάβουμε την κοινή αλληλευτική πολιτική στο γενικότερο ευρωπαϊκό ερευνητικό πλαίσιο. Εμείς πιστεύουμε ότι η αλία πρέπει να ξαναβρει τη θέση της στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα και να της δοθούν περισσότερα μέσα από ό,τι έχει τώρα. Κυρία Λοβίν, μιλήστε για 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλο ποσό. Μεν, αλλά έχουμε 27 κράτη-μέλη και η αλία δεν είναι μόνο θαλάσσια, είναι και εσωτερικών υδάτων. Εάν θέλουμε να εκπληρώσουμε όλες τις επιθυμίες όλων, τότε πολύ γρήγορα θα συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το ποσό των 6,5 δισεκατομμυρίων δεν φτάνει ούτε στο ένα εκατοστό του. Ο στόχος μας πρέπει να είναι, σε τελική ανάλυση, να χαράξουμε μια αλλιευτική πολιτική που για όλα τα... Που να προσέχει να υπάρχουν αρκετά αλληλευτικά αποθέματα, αρκετό εισόδημα και να είναι δίκαιοι και βιώσιμοι προς το περιβάλλον. Να Επίσης, πρέπει να δοθεί έμφαση στην αλληλεία μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή αλληλεία, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα τα τελευταία χρόνια με την εκβιομηχάνηση της αλληλείας. Επίσης, χρειαζόμαστε έναν ορισμό για την πλεονάζουσα αλληλευτική δυνατότητα. Πρέπει να έχουμε έναν ακριβή ορισμό και έχετε δίκιο που το αναφέρατε. Όμως, έχουμε ήδη ένα γενικό εύκολο ορισμό. Για παράδειγμα, οι ποσοστώσεις, όταν αυτές ξεπερνώνται, υπάρχει πλεόνασμα. Πρέπει να δούμε πώς θα τις ελέγξουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν σκάφη τα οποία υπεραλλιεύουν. Γεγονός είναι ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αν δεν το είχαμε, δεν θα, δεν θα κάναμε όλη αυτή τη συζήτηση. Τώρα, όσον αφορά την εμπειρία σας από την, τον διοικητικό τομέα και την μεταφορά αυτής από την ε, προηγούμενη στην επόμενη περίοδο. Έχετε δίκιο. Όταν, λέτε, όταν μιλάτε για πράγματα τα οποία μάθατε, πιστεύω αυτή η γνώση να μεταφερθεί και στα, άλλη, στα, και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη και στα νέα κράτη-μέλη όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Φυσικά και αυτά τα νέα κράτη-μέλη θα κάνουν λάθη και έχουν κάνει λάθη, όμως από τα λάθη μαθαίνουμε. Και εμείς εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε. Να δούμε πώς μπορούμε να εξαλείψουμε αυτά τα λάθη. Σε γενικές λοιπόν γραμμές, έλεγχος ναι, και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι συνειδητοποίησα στην επεξεργασία του κανονισμού ότι υπάρχουν πολλές χώλες που ακόμα δεν μας έχουν δώσει στατιστικά στοιχεία, στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε για να χαράξουμε μια συνετή πολιτική. Μας λείπουν στοιχεία λοιπόν σε πολλούς τομείς και ο έλεγχος για μένα είναι καταρχάς αρμοδιότητα των κρατών μελών, εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να αναλάβουμε και αυτό, αυτόν τον τομέα. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια. Δεδομένα λοιπόν, στατιστικά στοιχεία, δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά. Και παρακαλώ να υπάρξει στενή συνεργασία για τα δεδομένα αυτά ανάμεσα στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κούναστ. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον κύριο Καντέκ, να ακούσουμε και τον κύριο Γκάλαχερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που συνεισέφεραν στη συζήτηση το πρωί και μας διαφώτισαν σε σχέση με τα θέματα ειδικά των επιμέρους χωρών για αυτά που είπε η κυρία Ρόντουστ για την πλεονάζουσα δυνατότητα. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε αν μιλάμε για υπεραλίευση. Διότι η πλεονάζουσα δυνατότητα είναι κάτι που έχει αποτελέσει αιμονή για μας. Εάν υποθέσουμε ότι εγώ έχω μια βάρκα, ένα μεγάλο σκάφος, αλλά λίγο μόνο την ποσόστοση που μου αναλογεί, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος στις διάφορες χώρες στο παρελθόν όλοι μπορούσαμε να κατονομάσουμε επιμέρους χώρες που είχαν τέτοια προβλήματα, όμως δεν ξέρω τι συμβαίνει πλέον ακριβώς. Οι ποσοστώσεις, δεν ξέρω αν τηρούνται αυστηρά. Με το νέο λοιπόν αυτό ταμείο βλέπουμε να γίνεται λόγος για χρηματοδότηση ελέγχου και επιβολής των μέτρων. Εάν υπάρχει έλεγχο και επιβολή των μέτρων, θα έπρεπε να υπάρχουν τότε και κοινέ κυρώσει. Γιατί μιλάμε ιδάλω για κοινή αλλιευτική πολιτική. Κυρώσει και ποινέ που να είναι ίδιε σε όλη την Ευρώπη. Σε μερικέ χώρες ένα πλημέλημα μπορεί να θεωρείται κάπου ποινικό αδίκημα σε μια άλλη ή ε, διοικητικό παράπτωμα. Είναι λοιπόν σημαντικό το θέμα του ελέγχου και της ε, επιβολής. Νομίζω ότι ο έλεγχος εδώ είναι λοιπόν η απάντηση. Είναι σημαντικό να έχουμε το ταμείο αυτό των 6,5 δις, το οποίο να χρησιμοποιείται με σύνεση, αποτελεσματικά, αποδοτικά και να λαμβάνουν το κατάλληλο αντίτιμο και οι φορολογούμενοι που στηρίζουν το ταμείο αυτό. Και για την αλία και για την υδατοκαλλιέργεια. Εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε νομίζω περισσότερο στην υδατοκαλλιέργεια. Γιατί μπορούμε να την ελέγξουμε. Μπορούμε να ελέγξουμε το τι γίνεται, να προβλέψουμε και θέσεις εργασίας σε περιοχές που δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές πηγές απασχόλησης ή εκεί που έχουν αποδακατιστεί τα αλληλευτικά αποθέματα. Ενδεχομένω να υπάρχουν και υποδομέ που μπορούν να αξιοποιηθούν και να μην πάνε χαμένες. Εδώ έχουμε υπερβολικές ποσότητες φαριών που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγονται δηλαδή, και αυτό θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε ε, περισσότερο στην υδατοκαλλιέργεια. Εξίσου σημαντικό είναι η χρηματοδότηση να προβλεφθεί και για τεχνικά μέτρα συντήρησης. Διότι τα μέτρα αυτά δεν νομίζω να αρέσουν σε κανένα. Η απόρριψη δεν είναι κάτι νομίζω που βρίσκει κανένα σύμφωνο. Να λέμε τα ψάρια νέα, αλλά όχι για να τα πάμε πίσω στη θάλασσα μετά. Θα πρέπει λοιπόν περισσότερο κονδύλια να προβλεφθούν για την έρευνα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για στήριξη όλων των αποθεμάτων. Θέλουμε να περιοριστεί η θνησιμότητα, διότι από τη στιγμή που αλλιεύονται τα ψάρια, 99% ε, αποθνίσκουν. Μένουμε λοιπόν με τα χέρια άδεια. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε η έρευνα να μας οδηγήσει να χρησιμοποιούμε διαφορετικά είδη δικτυών, διαφορετικά μέτρα και με κάθε τρόπο να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά είναι οικολογικώς αξιόπιστα. Χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα μια βιώσιμη αλία ως ε, προστάτες ε, υπεύθυνοι των ε, αλληλευτικών αποθεμάτων πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτά θα υπάρχουν και στο μέλλον και για τις φώκες, δεν θέλω να επεκταθώ εδώ, αλλά οι περισσότεροι έχουμε υπόψη μας τις ε, φώκες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κατοικίδια. Όμως, κατοικέδια, Όμως στον Ατλαντικό οι φώκες είναι θηρευτικά και είναι πολύ επιθετικές. Άλλο τι γίνεται λοιπόν στη Βαλτική θάλασσα. Πρέπει να έρθετε να δείτε τι γίνεται στον Ατλαντικό ωκεανό. Αυτό βέβαια είναι συζήτηση για μια άλλη μέρα και μια ακόμη παρατήρηση όπως ακούστηκε στα πλαίσια του νέου ταμείου για την ανάπτυξη των λιμένων και τις υποδομές τους, θα πρέπει κάτι να προβλεφθεί. Ε, νομίζω όλοι όσοι γνωρίζουν τους μικρούς λιμένες ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουν ότι έχουν ε, αφανιστεί τα λιμάνια αυτά επειδή εξαρτώνταν από τα μικρά σκάφη και επειδή υπήρξε τέτοια πλέον υπερβολική αλίευση, στο, υπέρμετρη αλίευση στο παρελθόν. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν σε αυτά τα μικρά λιμάνια μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί, Γιατί ένα μικρό ποσοστό του ταμείου θα πρέπει να κατευθυνθεί ακριβώ για να εξυγχρονιστούν αυτοί οι μικροί λιμένε, να προβλεφθούν εγκαταστάσει. Εγκαταστάσει που να διευκολύνουν την ε, λιμένωση όχι τεράστιες μαρίνες ε, όπως αυτές που μπορεί να υπάρχουν σε άλλα μέρη της Ευρώπης, αλλά στη δική μου χώρα και αλλού, μικρά λιμανάκια ε, που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την επιβίωση και εκεί. Έχουν υποφέρει από ε, τη, τους κανόνες που επιβάλλουν τη χρήση συγκεκριμένων λιμένων. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει γενικότερη στήριξη, έστω και ένα μικρό ποσό, και τι προσφέρει μια μικρή ε, μαρίνα. Έστω ε, ε, κάποιες περιορισμένες εγκαταστάσεις. Κάπου να μπορεί να δέσει το σκάφος, να υπάρχουν δυνατότητες ε, να... Ε, λουτρών και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό και αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Πολλές ερωτήσεις έχουν τεθεί. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να τις δώσω παρόλα αυτά το λόγο για να παρέμβει. Κυρία Φλαμίνια. Καλημέρα σε όλους. Εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση Θάλασσας, τον τομέα που ασχολείται με τις ε, διευθυντικές πολιτικές. Τα τελευταία χρόνια ακριβώς ασχολούμαι με το θέμα του ταμείου, του αλληλευτικού ταμείου και της σημερινής πρότασης βέβαια για το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Θα ήθελα να καλύψω κάποια από τα ζητήματα που τέθηκαν, ιδίω ό,τι αφορά τον έλεγχο και τα συστήματα παρακολούθηση στο Ταμείο Θάλασσα και Αλίας. Και να δώσω και κάποιε διευκρινήσει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και το σύστημα διαχείριση, το μοντέλο μα. Δηλαδή τι τεχνικέ προδιαγραφέ που προβλέπει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη-μέλη. Εδώ να διευκρινίσω ότι όταν μιλάμε για έλεγχο, δεν μιλάμε για έλεγχο της αλίας. Έλεγχος και διαχείριση θα πει έλεγχος και διαχείριση των οικονομικών ροών. Θα πει συναλλαγές. Ε, μιλάμε για κάτι διαφορετικό λοιπόν από τον έλεγχο των αλλιευμάτων στα λιμάνια και το καθεξής. Να πω επίσης ότι το πρόβλημα προκύπτει από το περίπλοκο σύστημα της κοινή διαχείρισης. Η κοινή διαχείριση είναι μια πρακτική έκφραση της αρχής της επικουρικότητας. Εκεί αναγνωρίζουμε ότι σε επίπεδο κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις και να επιλέγονται οι χρηματοδοτούμενες ε, επιχειρήσεις. Αυτό έχει να κάνει πάλι με διαχείριση των κονδυλίων, ε, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδίδονται στα κράτη-μέλη και τα οποία έχουν ε, αρμόδιους οι οποίοι κανονίζουν πώ θα δαπανηθούν με, κάποιους, με γνώμονα κάποιου στόχου που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμω, αναγνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι οι αρμοδιότεροι προκειμένου να αποφασίσουν πού θα κατευθυνθούν τα κονδύλια αυτά. Η περιπλοκότητα τώρα από πού προκύπτει. Επειδή δίνουμε αποδίδουμε κονδύλια, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε και πού καταλήγουν. Τον έλεγχο όμω συνεχίζουν να τον έχουν τα κράτη-μέλη. Βεβαίω και είναι δύσκολο, βεβαίω και απαιτούνται πόροι, και προσπάθειες, όμως όποτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απευθυνθεί σε εξωτερικό συνεργάτη για έλεγχο, έχουν διαπιστωθεί ατασταλίες, παρατυπίες. Είναι λοιπόν σαν να μα λένε τα κράτη-μέλη ότι θέλουμε τα κονδύλια, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε και υπόλογοι και να λογοδοτούμε. Εντάξει, να παίρνετε τα κονδύλια και να έχετε την ελευθερία να αποφασίσετε πού θα τα επενδύσετε, αλλά πρέπει μετά να αναλαμβάνετε και την ευθύνη του να ελέγχετε το που πηγαίνουν τα κονδύλια αυτά. Ναι, είναι περίπλοκο, είναι ε, παθέ, αλλά είναι και απαραίτητο. Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι το δημόσιο χρήμα καταλήγει εκεί που πρέπει, εκεί που είχαμε αποφασίσει να το αποδώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο νομοθέτης έχει αποφασίσει ότι πρέπει να στηρίζουμε τους στόχους της κοινή αλληλευτικής πολιτικής όταν χρηματοδοτούμε κάτι βάσει του Ταμείου. Ένας από τους ομιλητές, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα όλων, έθεσε το θέμα του συστήματος της... Της διάλυσης. Εδώ αυτό μα θυμίζει ένα σύστημα που είχε να κάνει και με την απόσυρση των αυτοκινήτων, όπου δεν ξέραμε πού κατέληγαν τα διάφορα ποσά. Δεν θέλουμε να γίνει κάτι ανάλογο. Αυτό προκύπτει ε, δυστυχώ με το σύστημα κοινή διαχείριση. Είναι περίπλοκο. Προσπαθήσαμε με το νέο ταμείο να το απλοστέψουμε, συντονίζοντά το με τα υπόλοιπα ταμεία, όπω οι ε, επιδοτήσει που δεν θα δίνονται μέσω του νέου ταμείου. Δεν θα στηρίζονται λόγω χάρη εγκαταστάσεις των λιμένων μέσω του ταμείου αυτό, διότι αυτό μπορούν να το κάνουν ταμεία σε περιφερειακά επίπεδα που έχουν περισσότερη δυνατότητα και ευχέρεια οικονομική για να χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδου βελτιώσει. Όμω από το Ταμείο Θάλασσα και Αλία μπορούμε λόγω χάρη να χρηματοδοτήσουμε άλλα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σχέση με τους στόχους του στόχου όπω τον εξυγχρονισμό των λιμένων, των ίδιων λιμένων. Είμαστε βέβαιοι ότι με το συντονισμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Άλλο το τι χρηματοδοτεί το ταμείο αυτό, αλλά το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και με την επεξεργασία των προϊόντων που είναι πολύ διαφορετική από τις άλλους τομείς παραγωγής τροφίμων. Επενδύσεις λοιπόν που δεν θα πρέπει να επικαλύπτονται σε σχέση με τις δραστηριότητες άλλων ταμείων δεν σημαίνει ότι η επεξεργασία πια των ε, ψαριών δεν θα χρηματοδοτείται, απλώς θα χρηματοδοτείται από άλλες πηγές, άλλα ταμεία. Τώρα, για την ερμηνεία του κανονισμού. Αλήθεια είναι ότι κάπου υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν είναι πάντοτε απλό να ερμηνεύονται με ταχύτητα όλα τα σκέλη ενό νομοθετήματο αυτό. Όμω έχει να κάνει και με τον περίπλοκο χαρακτήρα του ίδιου του αλληλευτικού τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη ότι δεν μπορεί να αποδίδονται κονδύλια μόνο για διευθυντικού σκοπού. Πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι υπάρχουν και άλλοι στόχοι, όπω η προστασία των αποθεμάτων, η πλεονάζουσα δυνατότητα, η ικανότητα του σκάφου να αλλιεύει. Αυτά είναι έννοιε που δύσκολα μπορούν να, να γίνουν κατανοητέ σε άλλους τομείς. Εδώ απαιτείται, ναι, απαιτείται νομική μελέτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερμηνεύει όπου μπορεί, συνδυάζοντας και διαφορετικά στοιχεία. Την σαφή καθοδήγηση, γνωρίζοντα ότι σε επίπεδο κρατών μελών αποφασίζονται διάφορε επιχειρήσει και ενέργειε. Οπότε η εμπειρογνωμοσύνη χρειάζεται σε κάθε περίπτωση. Και από την άλλη, θέλουμε να διασφαλίσουμε τη μη διακριτική μεταχείριση των κρατών μελών μεταξύ του. Δηλαδή, ερμηνεύοντα. Μπορεί να καταλήξουμε σε μια προσπάθεια αρκετά επίπονη. Να σεβαστούμε ταυτόχρονα όλες αυτές τις αρχές. Σε ό,τι αφορά την αναδρομικότητα, να σας ε, βεβαιώσω ότι δεν είναι αυτή η αρχή που διέπει τι εργασίε τη Επιτροπή, η αναδρομικότητα. Έχει ληφθεί υπόψη μετά την έκδοση της έκθεσης του Ελεκτικού συνεδρίου για την πλεονάζουσα δυνατότητα. Και αν διαβάσετε την έκθεση αυτή θα συνειδητοποιήσετε πόσο δύσκολο ήταν να υλοποιηθεί, να εφαρμοστούν τα μέτρα και να υλοποιηθεί και η έννοια αυτή. Πραγματικά σε τέτοιες ε, περιπτώσεις τόσο ακραίες φαίνεται να χρειάζεται η αναδρομικότητα σε σχέση με τα πορίσματα και όλα τις έκθεσεις του Ελληνικού Συνεδρίου. Ελπίζω ότι αυτό σας δίνει μια εικόνα του πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα, ιδίως θα πρέπει να διαχειριστούμε ένα ταμείο με αυτή τη μέθοδο, τη μέθοδο της κοινή διαχείρισης. Όταν την παρακολούθηση την αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη και όταν τις περισσότερες αποφάσεις πρέπει να τις λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Ο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασκείται μόνον εξ post στις περισσότερες περιπτώσεις. Και δύο λόγια και για το Ταμείο θάλασσα και Αλίας. Δεν θέλω να μπω στι λεπτομέρειε, απλώ να διευκρινίσω ότι στην πρόταση από τα 17 άρθρα που αφορούν την Αλία υπάρχει μόνο μία διάταξη το άρθρο 32 που επιτρέπει τη δυνατότητα διαφοροποίηση. Το Ταμείο δεν επικεντρώνεται λοιπόν τη διαφοροποίηση των ε, δραστηριοτήτων. Τα 17 υπόλοιπα άρθρα ακριβώ αφορούν αποκλειστικώ και μόνο τον τομέα τη Αλία. Ωστόσο, αποφασίσαμε να μην αγνοήσουμε και την πραγματικότητα και εφόσον οι αλλιευτικέ δραστηριότητε σε κάποια μέρη της Ένωσης ε, όντως ε, περιορίζονται, σε αυτούς τους αλλιείς που θα αποφασίσουν να αλλάξουν επαγγελματικό κλάδο, θέλουμε να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος. Όχι, αυτά είχα να πω από τη δική μου πλευρά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Ευχαριστώ. Okay, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ολοκληρώνουμε το τμήμα αυτή τη συζήτηση και βλέπουμε, ε, κύριε Καντέκα, πώς θα εξασφαλίσουμε κονδύλια για να ε, σκοτώσουμε μερικές ε, φώκες και να φτιάξουμε μαρίνες. Εν συντομία θα ήθελα να πω ότι άκουσα κάποιες επικρίσεις από για το προηγούμενο ταμείο για την Ελία. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο το νέο Ταμείο Θάλασσας και να είναι πιο εύχριστο, πιο απλό και πιο διαφανές. Άκουσα και πολύ ενδιαφέροντα σχόλια που μερικές φορές συνάδουν με τις δικέ μου προτάσεις, αλλά άκουσα και κάποια μηνύματα, μερικά μάλιστα με θορύβησαν. Θα πρέπει, άπαξ παντός, να αποφύγουμε μία σύγχυση. Παρακαλώ κύριε Ρόντους, δώστε λίγη προσοχή. Εντάξει. Κύριε, Ρό... κύριε Ρόντουστ, είστε εισηγήτρια για το βασικό κανονισμό, οπότε θα ήθελα να με ακούσετε με προσοχή. Θα ήθελα άπαξ και διαπαντός να σταματήσει μία σύγχυση, να μην συγχαίουμε την αλληλευτική προσπάθεια με την, ικαν... ικανότητα. Η ικανότητα θεωρητικά αφορά την ισχύ σε κιλοβατόρες ενός σκάφους. Αυτή είναι η ικανότητα. Δεν υπάρχει σαφής ορισμός βέβαια αυτή τη στιγμή της ικανότητας, αλλά περί αυτού πρόκειται. Ενώ η αλλιευτική προσπάθεια είναι η ποσότητα των αλλιευμένων ε, ψαριών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ο κύριος Τραστόη πολύ σωστά μίλησε για τις ε, διαφορές της μετάφρασης μεταξύ της, αλλιευτικής, της ε, ικανότητας αλλιεύσης και της ικανότητας του σκάφους. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και μερικές φορές και στις μεταφράσεις υπάρχει σύγχυση. Όταν μιλούμε ικανότητα εννο, εννοούμε την ισχύ του πλοίου, του σκάφους και όχι την αλλιευτική, ε, τη δυνατότητα αλλίευσης του σκάφους. Γιατί ανάλογα με την ερμηνεία που θα υιοθετήσουμε καταλήγουμε σε διαφορετικό συμπέρασμα. Το απόγευμα θα γίνει συζήτηση και πάλι για το ΕΤΘΑ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όμως μας μίλησε με την γλωστή γλώσσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μεγάλη ευγλωτία, με ρητορική δυνότητα αλλά ουσιαστικά μία τρύπα στο νερό κάνατε. Είναι σαν να πνίξετε ψάρια, θα έλεγα, παραστατικά. Πολύ ωραία μας τα είπατε, αλλά απαντήσεις δεν μας δώσατε στους προβληματισμούς και τις απορίες μας. Αλλά θα επανέλθω μετά το δεύτερο πάνελ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Καντέκ. Θα ήθελα κατά το τέλος του δεύτερου πάνελ και το τέλος της συζήτησης να δώσω την ευκαιρία σε όλους τους καλεσμένους μας να ξαναλάβουν το λόγο για να σχολιάσουν ενδεχομένω ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Αλλά σε αυτή τη φάση θα προτιμούσα να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ, στο δεύτερο τμήμα της δημόσιας ακρόασης, που αφορά τις απόψεις των ενδιαφερομένων για τον νέο κανονισμό που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Ο πρώτος μας ομιλητής είναι ο κύριος Ζακ Βισόν, ο Διευθυντής της ε, Οργάνωσης Παραγωγών Αλιέων της Βρετάνης, θα ήθελα λοιπόν να του δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι διευθυντής μιας οργάνωσης παραγωγών με έδρα τη Βρετάνη. Ε, είναι η Αλής της Βρετάνης, μια οργάνωση ε, που καλύπτει 800 περίπου σκάφη με 100.000 τόνους ετησίως παραγωγής και έχει 300 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο. Μη ζητήσετε τη γνώμη μας για το ΕΤΘΑ. 107 αιτιολογικέ σκέψεις, 24 κεφάλαια, 154 άρθρα, 455 και μου δώσετε 10 λεπτά να μιλήσω για το ΕΤΘΑ. Είναι περίπλοκο λοιπόν το έργο και κολοσιαίο. Θα μπορούσαμε φυσικά να συνδυάσουμε τη συζήτηση αυτή με το βασικό κανονισμό. Είτε το κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς, γιατί το ΕΤΘΑ είναι ένα εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων του βασικού κανονισμού ουσιαστικά. Οπότε είναι αδύνατο κατά τη γνώμη μου μέσα σε 10 λεπτά να δώσω τις απόψεις μου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσης και Γι' αυτό εσκεμμένα θα επικεντρωθώ σε ένα από τα θέματα που αναφέρθηκε και το πρωί και αφορά τα αλληλευτικά δικαιώματα και τη διαχείρισή τους και πώς ε, θα παρέμβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας ε, και Αλίας προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της ελευτικής πολιτικής. Το ΕΤΘΑ λοιπόν είναι ένα νέο εργαλείο που θα πρέπει να θυγραμμίζεται και με το βασικό κανονισμό και με τον κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς. Γιατί αν είναι κακό ο βασικό κανονισμό και ο οργανισμό για την κοινή οργάνωση αγορά, θα είναι κακό και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία. Είναι συναφία αυτά τα θέματα και αλληλένδετα. Σε ό,τι αφορά τα αλληλευτικά δικαιώματα, Έχουμε ε, αφενός τα ατομικά δικαιώματα, αφετέρου τα συλλογικά δικαιώματα. Υπάρχει μια αντιπαράθεση. Ε, εγώ θα πάρω ως παράδειγμα την εξέλιξη της αλληλευτικής πίεσης και τη θνησιμότητα αλληλευτικών αποθεμάτων σε δύο βασικά αλληλευτικά είδη. Στο γάδο της Βορείου Θάλασσας που λίγο ή πολύ εμπίπτει σε διαχείριση με βάση τα ατομικά δικαιώματα γιατί η πολυ εμπιπτει διαχειριση με βαση τα χώρα η Νορβηγία που διαχειρίζεται το γάδο στηρίζεται στα ατομικά δικαιώματα και έχουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ε, ε βαλτικές χώρες ε, και έχουμε και το δεύτερο είδος ε, γάδου της Κελτικής θάλασσας με βασική, βασικές χώρες την Ιρλανδία και τη Γαλλία να εκμεταλλεύονται αυτά τα αλληλευτικά αποθέματα βλέπουμε ότι μετά τη θέση σε εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού από το 2002 έχουμε σαφή μείωση της θνησιμότητας ε, από λόγω, λόγω αλίας για το γάδο της Βορείου Θάλασσας, αλλά στη δεύτερη περίπτωση έχουμε αύξηση της θνησιμότητας και αυτό μας το λένε τα στοιχεία από του χρόνου, του 2013, θα φτάσουμε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση του ελευτικού αυτού αποθέματος. Οπότε η κατανομή ε, των ατομικών δικαιωμάτων δεν αποτελεί εγγύηση για τη συμμόρφωση με τους κανόνες. Και περίτρανη απόδειξη είναι ένα άρθρο του Fishing International γιατί η Ισλανδία που αναφέρεται πολύ συχνά ως ε, υπόδειγμα χώρας που έχει λύσει τα προβλήματά της με τα ατομικά δικαιώματα, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να έχει προβλήματα η Ισλανδία, γιατί υπάρχει μια μαύρη αγορά ε, ουσιαστικά για την υπόγλωσσα, για το αλληλευτικό είδος της υπόγλωσσας, οπότε θαυματουργή λύση δεν υπάρχει. Από τα δύο αυτά παραδείγματα, τι συμπεράσματα θα μπορούσαμε να αντλήσουμε. Καταρχήν, τα ατομικά δικαιώματα ε, λέει ένα κοινότυπο ότι ενισχύουν την υπεύθυνη στάση ενώ τα συλλογικά δικαιώματα ε, οδηγούν σε υπεραλίευση. Λάθος. Ε, δεν, ε, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Επίσης, η κατανομή των ατομικών συλλογικών δικαιωμάτων από μόνη της δεν ε, εγγυάται τη συμμόρφωση των κρατομελών με τους κανόνες, ούτε την επιτυχία της πολιτικής συντήρησης το κλειδί της επιτυχίας κατά τη γνώμη είναι ο τρόπος διαχείρισης των δικαιωμάτων. Οπότε και ο βασικός κανονισμός, αλλά και ο κανονισμός για την ΚΟΑ, αλλά και το θα μπορούν να συμβάλλουν σε μια αποτελεσματική πολιτική. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα γενικό πλαίσιο που αφορά τα δικαιώματα αλίευσης και που κατανέμει τις ε, μέγιστες αληφτικές ποσοστώσεις μεταξύ, με βάση μια κλίδα μεταξύ των κρατών μελών. Το γεγονός ότι μια χώρα έχει μια αλληλευτική ποσόστοση της επιτρέπει ε, να δώσει στους αλληλεί το δικαίωμα να αλλιεύσουν στα πλαίσια αυτής της ποσόστοσης και εν ανάγκη να προσαρμόσει στα, τον αλληλευτικό της στόλο στις ε, διαθέσιμες στα διαθέσιμα αλληλευτικά αποθέματα. Βέβαια δεν υπήρξε αυστηρή εφαρμογή παντού και το θέμα της εφαρμογής θα πρέπει να το βελτιώσουμε. Όταν έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης, κεντρικής διαχείρισης των ποσοστώσεων, τι συμβαίνει. Παρακολουθούμε καθημερινά την παραγωγή κάθε αλληλευτικού σκάφους και εφαρμόζουμε μέτρα που προσαρμόζονται σε κάθε αλληλευτικό στόλο, εξασφαλίζοντας και συμμόρφωση, παρακολουθώντας την εφαρμογή. Κάτι που είναι περίπλοκο όταν πρόκειται για μια συγκεκριμένη ποσόστοση. Γιατί ε, τα σκάφη δεν αλλιεύουν μόνο ένα αλλιευτικό είδος, αλλά πολύ, πολλά ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ένα αλλιευτικό ε, σκάφος ε, ε, αλλιεύει 100 τόνους γλώσσας, 17 τόνους αστακού, 6,7 γάδου ή μερλούκιο, συγγνώμη, και μάλιστα στην ίδια ζώνη, στη ζώνη 8. Βλέπετε το ίδιο σκάφος μέσα σε ένα χρόνο αλλιεύει πολλά διαφορετικά αλλιευτικά είδη. Οπότε είναι δύσκολο να γίνει η διαχείριση και ο έλεγχο μια ποσότητα. Ενώ κάθε χρόνο θα πρέπει να διαχειριστεί όχι μόνο ένα αλλιευτικό απόθεμα, μία ποσότητα αλλά πολύ περισσότερα ταυτόχρονα και να εξασφαλίσει έλεγχο και εφαρμογή. Υπάρχει δυσκολία λοιπόν και παρακολούθηση και διαχείριση, γιατί απομακρυνόμαστε από τη βάση. Οπότε τι συμβαίνει. Υπάρχει υπερκατανάλωση των ποσοστώσεων, κάτι που φυσικά είναι δυσάρεστο και μερικές φορές πρέπει να επιστρέψουμε το τμήμα της υπερκατανάλωσης. Το θέμα είναι ποιος είναι υπεύθυνο. Ε, το συγκεκριμένο ελευτικό σκάφος, ε, ποιος είναι ο υπεύθυνο για την επιστροφή. Και ως προς αυτό υπάρχει άγνοια. Για αποτελεσματική διαχείριση θα πρέπει να καθορίσουμε σαφείς κανόνες διαχείρισης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε ελευτικού στόλου και κάθε ελευτικού είδους θα πρέπει να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες όλων των αλληλευτικών σκαφών για να εξασφαλίσουμε συμμόρφωση με τους ε, κανόνες διαχείρισης, να μπορούμε να εντοπίζουμε ε, τους υπέτειους παραβίασης και να τους επιβάλλουμε άμεσα κυρώσεις και επίσης να εξασφαλίσουμε ε, προάσπιση των συμφερόντων όσων τηρούν τους κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε κοντά στους αλλήλει, κοντά στα σκάφη και να έχουμε κάποια κανονιστικά και οικονομικά μέσα στη διάθεσή μας για να ελοπίσουμε αυτούς τους στόχους. Ένα πιθανό μοντέλο θα ήταν αυτό που περιγράφω εδώ. Δηλαδή να προσδιορίσουμε ενδιάμεσα επίπεδα ευθύνη στη διαχείριση των δικαιωμάτων σε τοπικό επίπεδο που είναι και το πιο κατάλληλο. Για παράδειγμα με οργανώσεις παραγωγών που θα επιφορτίζονται και επίσημα με τη διαχείριση των δικαιωμάτων αλληλείας των μελών τους, είτε είναι αυτομικά αυτά είτε συλλογικά. Έτσι, το κράτος μέλος θα μπορούσε να εντοπίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν τοπικά και να επιφορτήσει κάθε τοπική οργάνωση να επιλύσει συγκεκριμένο πρόβλημα του συγκεκριμένου αλληλευτικού σκάφους ή συγκεκριμένης αλληλευτικής προσπάθειας. Υπάρχει ένας μηχανισμός ή προτείνεται ένας μηχανισμός για το σχέδιο παραγωγής και εμπορευματοποίησης του άρθρου 32 του κανονισμού για την ΚΟΑ. Είναι ένας μηχανισμός κατάλληλος για την ε, θέσπιση τέτοιων μέτρων λέει ότι ε, υποβάλλονται σε κάθε, εθνική, ε, σε κάθε εθνική αρχή ένα σχέδιο ε, παραγωγής και εμπορευματοποίηση προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του άρθρου 3. Το άρθρο 3 είναι το αντίστοιχο ε, της, ε, το άρθρο υλοποίηση των γενικών στόχων της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Τι λείπει. Λείπει διαφάνεια, γιατί για να υπάρχει διαφάνεια χρειαζόμαστε κοινού. Κανόνε διαχείριση. Ο κύριο Γκάλεχερ πολύ σωστά είπε ότι θα πρέπει και οι κυρώσει να είναι κοινέ και εναρμονισμένε, αλλά και οι κανόνε διαχείριση να είναι κοινοί, ώστε να έχουν όλοι στην Ευρώπη εμπιστοσύνη στην ε, εφαρμογή των κανόνων και στην τήρηση του νόμου. Το σχέδιο παραγωγή ε, και εμπορευματοποίηση, το άρθρο 32 τη ΣΚΟΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει ένα σημαντικό σκέλο που αφορά τη διαχείριση των αναλευτικών δικαιωμάτων των μελών. Η δυσκολία στην ισχύουσα ΚΟΑ έγκυται στο ότι το περιεχόμενο των σχεδίων αυτών παραγωγής και εμπαρευματοποίησης ε, ε, προβλέπει να καθορίζεται από κατεξουδιώδηση πράξης με βάση το άρθρο 33 της ΚΟΑ. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να γίνει σε πολιτικό συζή... επίπεδο συζήτηση για το περιεχόμενο αυτών των σχεδίων παραγωγής και παρευματοποίηση και να αναφέρεται και στο βασικό κανονισμό. Επίσης, ε, θα πρέπει οι διαχειριστές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να τροποποιηθεί το άρθρο 7 του σχεδίου για την κοινή οργάνωση αγοράς προκειμένου να υπάρχει μια εντολή διαχείρισης των αλληλευτικών δικαιωμάτων, κάτι που δεν υπάρχει. Στο άρθρο 8 της ΚΟΑ θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στους αρμόδιους για τη διαχείριση φορείς και να προσθεθεί ένα εδάφιο το εδάφιο G, για παράδειγμα, που να λέει επιβάλλονται κυρώσει στα μέλη που δεν δε συμμορφώνονται με τους στόχους που περιλαμβάνει το σχέδιο παραγωγής και εμπορευματοποίησης. Επίσης, σε ό,τι αφορά την κοινή οργάνωση αγοράς, λείπει και ένα άρθρο 19, γιατί προβλέπεται μια ανάκληση της αναγνώρισης σε περίπτωση έλλειψης σχεδίου ε, παραγωγής και εμπορευματοποίησης ή α, ε, λόγω παραβίασης των εφαρμοστικών κανόνων θα πρέπει όταν δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες ε, να διαγράφονται ε, τελείως αυτές οι οργανώσεις. Σε ό,τι αφορά το ΕΤΘΑ, θα πρέπει το ΕΤΘΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και να στηρίζει άμεσα την προετοιμασία και την εφαρμογή των σχεδίων και να μην είναι προαιρετικό κάτι τέτοιο, να γίνεται συστηματικά. Τώρα, κάποιε λεπτομέρειε να τροποποιηθεί η τελική σκέψη 62 του ΕΤΘΑ, γιατί είναι αντιφατικό αντιφατική με το επόμενο κείμενο. Επίσης, στο άρθρο 15 του ΕΤΘΑ προβλέπονται ε, χρηματοδοτήσεις, αλλά νομίζω ότι ε, συντακτικά υπάρχει πρόβλημα. Εκεί θα πρέπει να διορθωθεί η διατύπωση. Έχω ξεπεράσει λίγο το χρόνο μου. Θα ήθελα να κατακλείδη να επανέλθω ε, ε, στη θνησιμότητα του γάδου της Κελτικής ε, θάλασσας, ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα με βάση τον ισχύοντα κανονισμό περάσαμε από ένα επίπεδο θρησιμότητας 0,5 πάνω από το FMSY σε ένα ποσοστό που το 2010, τέλη 2010, ήταν 0,1 πάνω από το FMSY. Δηλαδή φτάσαμε στην μέγιστη, θα φτάσουμε στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση στα τέλη του έτους. Αυτές είναι οι προβλέψεις μας. Τώρα, πώς καταλήξαμε στο αποτέλεσμα αυτό. Ε, πολύ θεαματική η κατάσταση αυτού του ελευτικού αποθέματος. Το 2003 οι οργανώσεις παραγωγών, οι ενδιαφερόμενες από το ελευτικό αυτό, απο, αυτό αυτο κυρίως α, ε, Ιρλανδικές, α, ε, με, ε, μ, με διάφορες Ιρλανδικές οργανώσεις, η FPO, CAIFO και οργανώσεις της Βρετάνης, Μπροστά στην ενισχυτική κατάσταση του αποθέματος γάδου, προτείναμε κάποια μέτρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γάδο τη Κελτικής ε, θάλασσα και κάθε χρόνο για δύο μήνες ε, βλέπετε τα, στα παραλληλόγραμμα αυτά απαγορεύεται αλίευση. Έκτοτε έχει μειωθεί η θνησιμότητα, ανασυγκροτούνται τα αλλιευτικά αποθέματα και περάσαμε πια την κρίσιμη βιομάζα, τη βιομάζα ε, προφύλαξης. Και επιτύχαμε την ανατροπή αυτής της αρνητικής τάσης χάρη στη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων ε, παραγωγών. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Μου δίνετε ακόμη ένα λεπτάκι για να σας παρουσιάσω μία διαφάνεια για τα σχέδια της ε, διάλυσης ή ε, αποχώρησης των αλλιών από την ελευτική προσπάθεια και πάλι για το γάδο της Κελτικής. Έχετε το επίπεδο της βιομάζας στην πράσινη καμπύλη ενώ στα, στις μπλε στήλες έχουμε τον αριθμό των σκαφών που αλλιεύουν στο αλλιευτικό αυτό απόθεμα. Από το 2005 στη Γαλλία εφαρμόσαμε κάποια στοχευμένα σχέδια για τα σκάφη που είχαν εθνικές άδειες που ζητούν δικαίωμα πρόσβασης στην εκμετάλλευση αυτών των αποθεμάτων. Και βλέπετε ότι ήταν μικρό ο αντίκτυπο στο στόλο το 2005 και το 2006, πιο σημαντικός 2007 και 2008, το κόκκινο σημείο τη στήλη. Εκεί έχουμε τα σκάφη που ε, εξήλθαν από το στόλο. Και μάλιστα κάναμε μια προσωμείωση για να δούμε πού ε, θα έφτανε η βιομάζα αυτών των αποθεμάτων αν δεν είχαν ε, ε, δεν είχαν εξέλθει ορισμένα πλοία από το σκάφο. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχαμε ανακτήσει τη βιομάζα αν είχαν παραμείνει όλα τα ελευτικά σκάφη στο στόλο. Μπορούμε να έχουμε μια γενική εντύπωση για τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα αυτού του μέτρου, εξόδου από τον ελευτικό στόλο κάποιων πλοίων. Αν είναι όμως στοχευμένα αυτά τα σχέδια και σε συγκεκριμένες υδατινές λεκάνες, όπως σε ε, ένα συγκεκριμένο απόθεμα, με συνεργασία των ε, χωρών, ώστε να γίνει ένα τέτοιο σχέδιο διάλυσης ή εξόδου από τον ελευτικό στόλο, συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου Γαλλίας εν προκειμένου, πραγματικά τότε θα έχουμε μια πολύ θετική επίδραση. Ευχαριστούμε κύριε Πισού. Ο κύριος Αλμπερίκο Σεμιόλη τώρα, από την Λέγα Κοπ, για την αλία στην Καμπανία. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας και σας Πρόεδρε για αυτή την ευκαιρία. Είμαι εκπρόσωπος μιας ε, ένωσης αλίας αλλά και εγώ ψαρεύω ο ίδιος. Είμαι εκπρόσωπος λοιπόν της μικρής παράκτειας αλίας. Στόχος μου είναι να σας εκφράσω λοιπόν την καθημερινή μας εμπειρία από τη θάλασσα. Η σημερινή μου παρουσίαση θέλει να δώσω την άποψη λοιπόν της μικρής παράκτειας αλίας σε σχέση με το νέο Ταμείο για τα θαλάσσια ζητήματα και την αλία. Προτού σταθώ στα βασικά ζητήματα του Ταμείου, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα ήθελα να κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις διότι θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε και υπό το φως των όσο σήμερα ακούσαμε σε σχέση με τον έλεγχο. Ενώ η Επιτροπή με τους κανονισμούς της σε σχέση με την επαγγελματική αλία έχει καθορίσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, η Ιταλία και η Καμπανία λόγου χάρη ε, ταξιδεύει και να ψηπλοεί σε ένα διαφορετικό ημισφαίριο, σε ένα διαφορετικό κόσμο. Όλοι οι προηγούμενοι κανονισμοί, όπως ο δημοσιονομικός κανονισμός για την αλία, και το Ταμείο Αλίας κάνουν μια προσπάθεια να ελέγχεται η μικρή κλίμακα παράκτη αλία. Όμως, ενώ εγκαινιάζονται κοινοτικέ πολιτικές για αυτόν τον τομέα, οι ίδιες οι κοινοτικέ πολιτικές στην πράξη δεν λαμβάνουν υπόψη κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις. Να δώσω κάποια παραδείγματα. Στο παρελθόν, η παράκτη αλία μικρής κλίμακας συνήθως ε, υλοποιούνταν με συγκεκριμένα σκάφη μεγάλου όγκου που, που ήταν είτε τετράτες είτε γρηγροί. Σήμερα με τον έλεγχο της ε, παράκτιας ηλίας μικρής κλίμακας φαίνεται να εφαρμόζονται σωστά όσα προβλέπονται από τον ελληνικό κανονισμό. Περίεργο βέβαια αυτό ερχόμενο από την κατεύθυνση ενός ε, ψαρά. Όμω, ενώ φαίνεται τώρα να πηγαίνουν καλά ακριβώ για την επαγγελματική αλεία, από μια άλλη άποψη πάνε πολύ άσχημα. Σήμερα, οι αλεί παράκτεια ε, μικρή κλίμακα αλεία έχουν κάποιο μεγάλο ανταγωνιστή. Του ερασιτέχνε αλλοί. Ενώ λοιπόν οι κοινοτικοί κανονισμοί πολύ καλά έχει διευθετήσει, έχει απαγορεύσει όσα δεν πρέπει να γίνονται στην επαγγελματική αλεία, το άρθρο 17 μόλις γίνεται λόγος για την ερασιτεχνική αλία. Έτσι, σήμερα στην Ιταλία έχουμε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ερασιτέχνες αλίες που βγαίνουν στη θάλασσα χωρίς κανένα είδους άδεια, κανόνα. Και κανέναν έλεγχο. Είναι αδύνατο να ελεγχθούν οι ερασιτέχνε αλίες. Δεν είναι γνωστά τα σκάφα, δεν υπάρχουν ε, μητρώα, δεν ε, καταγράφονται, δεν γίνεται τίποτα στην περίπτωση τη ερασιτεχνική αλίας, όπω για την επαγγελματική. Έτσι, η Ιταλική νομοθεσία για την ε, εραστεχνική αλεία έχει μείνει στους κανόνες που προβλέπονταν το 55. Ε, έτσι λοιπόν, να δώσω το παράδειγμα ειδών όπως ε, ο κέφαλας, το περιγράφει αυτό και το γραπτό μου κείμενο, αλλά θα ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ψαρεύονται τέτοια ψάρια όπως οι κεφαλάδες. Τα μικρά αυτά σκάφη των ερασιτεχνών ε, ψαράδων δεν τείνουν να ανοίγονται πολύ στο πέλαγος. Ψαρεύουν λοιπόν ε, τα προϊόντα αυτά, τα ψάρια αυτά και τα εμπορεύονται καταπευθεία στα εστιατόρια και τους αγοραστές. Βεβαίω, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό το ερυθρού τόνου, ο οποίο στην ε, καμπανία άγγιζε επίπεδα ρεκόρ. 49 σκάφη σε όλη την Ιταλία, 12 πλέον με τους νέους κανόνες, 7 συγκεκριμένα στην καμπανία. Καλό αυτό, είναι καλός ο έλεγχος και το 11, το 2011 1.600 σκάφη είχαν έγκριση ερασιτεχνικής αλίας από το Υπουργείο Γεωργίας και Αλληλευτικών Ζητημάτων. Ακόμα και τώρα οι ερασιτέχνες αλείς θα ψαρεύουν και θα ξεπερνούν τις ποσοστώσεις, τα όρια των ποσοστώσεων του 2011 που είναι πλέον στα επίπεδα του 35%. Γιατί ακριβώς δεν ελέγχονται. Και για άλλα από όπως οι σφυρίδες, ε, οι συναγρίδες και τα μαγιάτικα είναι ακριβώς αλλιεύματα αποκλειστικά της ερασιτεχνικής αλίας, οι οποίοι ψαρεύουν με ζωντανά δολώματα. Και αυτό βεβαίως πλήττει τα αποθέματα. Άρα Εάν θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την ε, παράκτη αλία μικρή κλίμακα και το ταμείο, θα πρέπει να σκεφτούμε, να δούμε ακριβώ τι έγινε στην ε, καμπανία. Όχι, δεν εμπόδισαν οι κανόνες του άρθρου 27 και ο περιορισμός του αριθμού των σκαφών. Όχι, οι αλλοίες απλώς έχουν γίνει ερασιτέχνες. Η ερασιτεχνική αλία με κανέναν τρόπο δεν ελέγχεται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει μια σειρά από κανόνες αυστηρούς που απαγορεύουν ένα σωρό πράγματα, όπως για τον ερυθρό τόνο, που προβλέπει και συγκεκριμένες μεθόδους αλίευσης λόγου χάρη, για τον ισοπαγγελματίας αλληλής αλλά όχι για τους ερασιτέχνες. Εδώ να θυμηθούμε ότι αυτά είναι γνωστά και με τον Υπουργό που είχαμε πρόσφατα, ο οποίος ήταν ε, φανατικός ψαράς ε, της ρασιτεχνικής αλίας που συζητάμε. Άρα, ωραία είναι η έλεγχη, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό το φαινόμενο πρέπει να του δοθεί ιδέουσα προσοχή. Διότι το τι θα συμβεί από τώρα ως την έγκριση του κανονισμού για το Ταμείο είναι γνωστό. Μέχρι τώρα, πέραν από τα κονδύλια που απευθύνονταν στον εξυγχρονισμό, ε, κάποια αποδίδονταν και στην ε, έξοδο κάποιων σκαφών από τον αλληλευτικό στόλο, αλλά δεν έχουν να κάνουν με την αριστεχνική αλεία. Ας υποθέσουμε ότι επί 20 χρόνια την βάρκα που χρησιμοποίησα για να τεχνική αλεία δεν την έλεγξε κανείς. Οι έλεγχοι θα γίνουν μόνο από τη στιγμή που αρχίζουν να λειτουργούν οι κανόνες, χωρίς να αλλάξει το είδος και η μέθοδος αλίας. Εδώ ελπίζω να ακούει αυτά που λέω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τα έχω πει από όλα τα δυνατά βήματα, αλλά καλό θα ήταν να, ε, να ακούγεται και η φωνή της μικρής αλίας. Ίσως να μας ακούνε ακριβώς γιατί είμαστε μικροί. Όμως, ο κανονισμός αυτός είναι αυστηρός και θα πρέπει να είναι αυστηρός για τον περιορισμό της αεραστεχνικής αλίας. Διότι εάν εν τέλει αξιολογηθούν τα αποθέματα με τον έλεγχο, ε, με τον εφαρμογή των μέτρων, θα πρέπει να δούμε εάν περιορίστηκε η κατάρρευση των αποθεμάτων και τι γίνεται και με τη θνησιμότητα. Φαίνεται ότι η πλεονάζουσα αλίευση όμω οφείλεται στου επαγγελματίε αλίε και όχι στου ερασιτέχνε. Και α υποθέσουμε ότι ο κανονισμό διευθετεί τελικά και την ερασιτεχνική αλία με τρόπο αυστηρό. Α υποθέσουμε ότι και για του ερασιτέχνε αλίες προβλέπονταν οι ίδιε κυρώσει που προβλέπονται για του επαγγελματίε. Μου φαίνεται αστείο ότι για μια σοβαρή παράβαση, αλίευση ενό ερυθνού τόνου λόγου χάρη, ο επαγγελματία ψαρά δεν έχει πρόσβαση στα κονδύλια, ενώ οι εραστέχνε δεν έχουν καμία, κανένα περιορισμό. Μία διοικητική μόνο κύρωση. Φανταστείτε λοιπόν πόσο του νοιάζει όλο αυτό του εραστέχνε αλείς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι λειτουργήσε και τι πήγε καλά με το Ταμείο Αλίας και τι θα πρέπει να αλλάξει στο Ταμείο Θαλασσίων Ζητημάτων και Αλίας. Είναι πολλοί οι φορεί που εμπλέκονται στη διαχείριση του Ταμείου. Οι φορεί τουλάχιστον στην Καπανία, τοπικού επίπεδου δηλαδή, έχουν συνεργαστεί καλά, διότι ε, έτσι οι είναι και πιο κοντά στους φορείς πληρωμής. Όμως, τα κέντρα πληρωμής με τους περίπλοκους χάρους που προβλέπονται, κάποιε φορέ καθυστερούν πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν επίτροπες, το κράτος, οι περιφέρειες, οι φορεί τοπικής αυτοδιοίκηση, είναι πολλοί φορείς που εμπλέκονται. Πρέπει όμως εδώ να πούμε ότι πολλές από τις δραστηριότητε που έχουν εκχωρηθεί Πολλά από τα μέτρα που έχουν ε, ε, εκχωρηθεί, ανατεθεί στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως οι ομάδες ε, παράκτητες δράσης, είναι στοιχεία που τόσο δεν θα μπορούσαν να ελεγχθούν σε κεντρικό επίπεδο. Οι περιφερειακές λοιπόν οργανώσεις έχουν καθοριστικότερο ρόλο στο πώς θα υλοποιηθούν τα μέτρα του νέου ταμείου. Τώρα, για το άρθρο 26 και 27 του κανονισμού του κανονισμού 1198 του 2006. Εδώ δεν ε, είναι επαρκή τα μέτρα που προβλέπονται, ιδίως για τους μεμονωμένους αλληλείς σε τοπικό επίπεδο. Στην Ιταλία έχουμε συνεταιρισμού αλλιέων με 400 μέλη πολλές φορές, με 200 σκάφη. Ο νέος λοιπόν κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει και τη δυνατότητα εκπροσώπησης ομάδων αλλίων, όχι μόνο εξατομικευμένων αλλίων, που στην Ιταλία δεν υπάρχει σε φορολογικό επίπεδο. Επίσης, το άρθρο 37 στο εδάφιο M θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η ευκαιρία, αλλά στην Ιταλία που έχει ήδη ακολουθήσει μια οδό αυτήν της ταύτισης των τοπικών ε, προγραμμάτων διαχείρισης ε, του 37M με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό 1967 τελικά οδηγούν σε περίπλοκα μέτρα. Δηλαδή ζητάμε από τους αλληλείς να προβλέψουν ένα πρότυπο σχεδίου δράσης ε, όπως ορίζεται από τον κανονισμό 1967. Τώρα στο άρθρο 37 αναφέρονται τα συλλογικά δικαιώματα εδώ θα μπορούσαμε να βρούμε μια ευκαιρία για το μέλλον. Δηλαδή, εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει περαιτέρω αυτούς τους προβληματισμούς. Τώρα, η εμπειρία μας από τις ομάδες δράσης στην παράκτια Αλία, η ίδια δηλαδή η πείρα της Αλίας σε καθημερινό επίπεδο, δείχνει ότι συμμετέχουν ιδιαίτερος και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα μέλη. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Ε, αυτό είναι το σημαντικό από την πλευρά των αλλίων. Για το Ταμείο λοιπόν Θαλασσίων Ζητημάτων και Αλία έχουν υποθεί ήδη πάρα πολλά. Θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου. Απλώ να υπάρχει δυνατότητα για χρηματοδότηση όσο να έχουν ε, διαπράξει σοβαρά παραπτώματα. Αυτό ε, ξανανοίγει μια συζήτηση για το τι είναι σοβαρό παράπτωμα σε κάθε χώρα και πώ αντιλαμβάνονται τα διάφορα κάτι μέλη. Δηλαδή, κάπου ε, μπορεί να είναι η χρήση συγκεκριμένων αλληλευτικών μεθόδων σε κάποιες ε, περιπτώσεις για την Ιταλία, για άλλους μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Επίσης, ο τουρισμός ε, για αλληλευτικούς σκοπούς είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και κάτι που έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη και ενδιαφέρει πολύ τους αλείς σε τουριστικές μάλιστα ζώνες. Στην ε, Ιταλία έχουμε πάλι εδώ συνεταιρισμούς. Το 50.000 ευρώ προβλέπεται ως μέγιστη δαπάνη, ως ποσό μέγιστης δαπάνης, για την οικονομική συνδρομή στο 50% του ισολογισμού του, της επιχείρησης. Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν τουλάχιστον 400, 400 μέλη. Επίσης, για την οριστική πάυση δραστηριοτήτων, εδώ τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι πολύ σοβαρά, διότι η εμπειρία μας από τα προγράμματα διαχείρισης έχουν δείξει στην καμπανία τουλάχιστον ότι είναι δύσκολο να υλοποιηθούν όλα αυτά τα στοιχεία για την μικρή αλία. Στην ε, καμπανία η ομάδα αλίας ε, που δεν ήταν ε, και γνωστή δεν μπόρεσε τελικά να στηριχθεί από αυτή τη διαδικασία και στην Ιταλία σήμερα υπάρχει μόνος ένας αλιέας ο οποίος ε, στηρίχθηκε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε κύριε Σεμιολή. Ευχαριστώ κύριε Σεμιολή. Βλέπω ότι συναντάβεστε από έναν εκπρόσωπο της αλίας μικρής κλίμακας. Περνάμε στον επόμενο μιλητή, που είναι ο κύριος Βαυζίνιετς Βαυζίνιακ, συγγνώμη για την προφορά, λέει ο πρόεδρος, που είναι βασικό σύμβουλος της Πολωνικής Ένωσης Αλλιέων για, την κοινή, για τη μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Παρακαλώ κύριε Βαυζίνιακ, έχετε το λόγο. Αξιότιμη κυρίε και κύριοι, κύριε πρόεδρε, Ονομάζομαι Βαυζίνιες Βαυζίνιας και είμαι καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Στσέτσιν. Θα σας παρουσιάσω τη θέση των Πολωνών Αλλιέων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της αλλιείας στην Βαλτική θάλασσα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα όμως να ευχαριστήσω ε, εκ μέρους των Αλλιέων την Επιτροπή σας για την οργάνωση της δημόσιας ακρόσης. Η θέση που θα σας παρουσιάσω είναι αποτέλεσμα διαβούλευση με ολόκληρο το φάσμα των ε, Πολωνών Αλλιέων. Στόχος της διαβούλευσης ήταν η διαμόρφωση της κοινή θέση των Αλλιέων σε ό,τι αφορά μια αηφόρο διαχείριση τη αλίας στη Βαλτική και ιδιαίτερα στα χωρικά ύδατα της Πολωνία. Οι Πολωνοί αλλοί στάσσονται υπέρ μια αηφόρου διαχείρισης της αλίας σε όλε τι υδάτινε λεκάνε, θάλασσε, ωκεανού και ιδιαίτερα στη Βαλτική, γιατί ε, την ε, Βαλτική εκμεταλλεύονται μαζί με άλλε Βαλτικέ χώρε. Οι απόψει του, ε, μάλιστα περιλαμβάνονται στον Πολωνικό Κώδικα υπεύθυνη Αλίας. Μία υφόρος διαχείριση τη αλίας ε, μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με περιφερειακή διαχείριση δάτινων λεκανών και θαλασσών. Γιατί κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα τα ύδατα από εκείνους που ζουν και εργάζονται στι όχθε του. Οι Πολωνοί ε, αλληλείς έχουν ζωηρό ενδιαφέρον για μια ορθολογική διαχείριση των ε, αποθεμάτων του γάδου της ε, Βαλτικής και ιδιαίτερα του κόλπου του Γκτάνσκ, κάτι που σχετίζεται με τη συνεργασία με τους αλληλείς των γειτονικών χωρών. Είμαστε υπέρ του ψηφίσματος της, του Δευτέρας Απριλίου του 2012 για άκρηση του κανονισμού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου 2012-0077 για την αναθεώρηση του κανονισμού 1098-2007 που προβλέπει μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου ε, στη Βαλτική και την αλία των αποθεμάτων αυτών. Σε ό,τι αφορά ε, την ελαστική διαχείριση της πολιτικής ε, που θα προσαρμόζει το νομικό καθεστώς στα επιστημονικά πορίσματα σε ό,τι αφορά την αλλαγή της κατάστασης του αποθέματος. Είμαστε εκεί υπέρ της ορθολογικής διαχείρισης των αποθεμάτων ε, ε, αρινής και φθινοπορεινής ρέγγας που φτάνουν στις πολωνικές ε, και σουηδικές ακτές και είμαστε υπέρ της προστασίας των τόπων αναπαραγωγής και τη σωστή ανάπτυξη των ηχθιδίων της ρέγγας. Είμαστε υπέρ ορθολογικής διαχείρισης και των αποθεμάτων σαρδελόρεγγας, σολομού και επίπεδων ψαριών και είμαστε με Σουηδούς κυρίως και Δανούς αλείς. Οι Πολωνοί ε, αλληλεί είναι κατά των αλλιευμάτων για παρασκευή χθιαλεύρων, τουλάχιστον είναι υπέρ του περιορισμού, γιατί τέτοιου είδου ε, αλληλεία απειλεί το οικοσύστημα των ζωντανών αποθεμάτων στη Βαλτική. Η ανεπιφύλακτη συμφωνία για τέτοιου είδου ε, αλλίευση διαταράσσει την αηφόρο αλληλεία στη Βαλτική γιατί επηρεάζει την ισορροπία μεταξύ των αλλιευτικών ειδών που διαβίουν στη Βαλτική και οδηγούν σε υπεραλίευση. Η Βαλτική είναι πολύ μικρή θάλασσα για να μην έχει σημασία τέτοια αλία στη γενική κατάσταση των αποθεμάτων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να, να περιοριστεί η παραλίευση ιδιαίτερα σαρδελόρεγγας ε, και ρέγγας ε, και να γίνει σωστή διάκριση μεταξύ της αλίευσης για καταναλωτικούς στόχους και για την παρασκευή ε, ή ηχθιαλεύρων. Ε, μία εναλλακτική λύση για την αλία θα ήταν η διαχείριση των παραλιευμάτων προκειμένου να μην απορρίπτονται τα νεκρά ψάρια στη θάλασσα. Θα πρέπει επίση να γίνει μία σωστή διαχείριση ανάλογα με τον προορισμό ε, για την κατανάλωση ή για την παραγωγή ζωοτροφών. Θα πρέπει να λυθούν κάποια τεχνικά και οικονομικά μέτρα για το πρόβλημα αυτό. Γιατί αν θεωρηθούν τυχαία ακούσει αυτά τα παραλιεύματα και περιλαμβάνοντα το ημερολόγιο πλοίου ή στα έγγραφα τη πρώτη πληρωμή, θα είχαμε την ευκαιρία για έναν αυτόματο αυτοέλεγχο της αλίευσης, κάτι που θα μπορεί να χρησιμοποιεί είτε το κράτος είτε η Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης για να διενεργήσει έλεγχο των αλιευμάτων και των αποθεμάτων. Επίσης, ε, τα παραλιεύματα θα πρέπει να μεταφέρονται στα λιμάνια από τους αλίες που τα έχουν αλιεύσει. Κύριε Βαυζίνη, μήπως θα μπορούσατε να επιβραδύνετε λίγο το αριθμό σας, γιατί πραγματικά μιλάτε με ηλικιώδη ταχύτητα. Παρακαλώ, αφού διαβάσετε το κείμενό σας, τουλάχιστον κάντε το με πιο αργό τρόπο. Μία υφόρος ε, διαχείριση της αλίας στηρίζεται και στην ε, προστασία των θηλαστικών και των θαλάσσιων πτηνών. Μια ανθρωπιστική προσέγγιση στο θέμα αυτό αφορά μια ε, εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων ειδών η συνεργασία όλων των αλλιών της ε, Βαλτικής θάλασσας ε, θα πρέπει να εξασφαλίσει μια ισορροπημένη διαταραχή και όχι μια υπερβολική ανάπτυξη ενός είδους εις βάρος των άλλων. Για παράδειγμα έχουμε τον Κορμοράνο ε, και συνεργασία μεταξύ των αλλιών της Βαλτικής σε θέματα κορμοράνου και φαιάς φώκες που είναι θηρευτές που απειλούν την τοπική αλεία. Σε ό,τι αφορά τα αλευτικά εργαλεία, η Πολωνία Αλίας είναι υπέρ της διατήρηση των ισχυών των αλευτικών εργαλείων στην Βαλτική και είμαστε υπέρ της επαναχρησιμοποίησης των παρασυρώμενων δικτυών. Γιατί η απαγόρευσή του στηρίχθηκε στην υποτιθέμενη προστασία του μαρσουίνου, τη φώκε μαρσουίνου. Αλλά τα, τα παρασυρώμενα δικτύα χρησιμοποιούνται εκεί που δεν υπάρχουν μαρσουίνοι. Θα πρέπει επίσης ε, να δημιουργηθούν ε, και μέτρα για να ε, προστατευτούν θηλαστικά και πτηνά από την εμπλοκή τους σε τέτοια δίχτυα. Η παγκόσμια κρίση της αλίας ε, προβληματίζει και τους Πολωνούς ε, αλείς που ενδιαφέρονται για την διατήρηση των αλληλευτικών αποθευμάτων και μια υφόρο αλία που να επιτρέπει την αυτοανανέωση των αποθεμάτων σε θάλασσες, ωκεανούς και ιδιαίτερα στην, Βαλτική προκειμένου να εξασφαλιστεί η φόρος εκμετάλλευση. Επίσης ε, ζητούν δίκαιη μεταχείριση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ίσους όρους με τους υπόλοιπους αλίες, γιατί είναι άδικη μερικές φορές η μεταχείριση των πολωνών αλίων. Υπάρχουν ενισχυμένοι έλεγχοι των εκφορτώσεων, ενώ πολωνοί επιθεωρητές δεν μπορούν να ελέγξουν πλοία άλλων σημαίων, ιδιαίτερα μεγάλες μηχανότρατες. Επίσης ε, υπάρχει μια έλλειψη ελαστικότητας ό,τι αφορά τη λήψη, <coughs> συγγνώμη, τη λήψη υπόψη των διακαίνων δικτύων ΤΑΦ 90 ή Μπακόμα. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στον κανονισμό 2011-0380. Αναφέρεται στο 2793. Οι προκαταβολέ σε επίπεδο 4% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία θα πρέπει να συμβάλλουν στην επιτάχυση τη διαδικασία εφαρμογή του λειτουργικού προγράμματο. Ένα τόσο χαμηλό όμω ποσοστό προκαταβολή δεν μπορεί να επισπεύσει την εφαρμογή του προγράμματο. ιδιαίτερα όταν οι δόσει είναι 2% πιο πιθανή βοήθεια προκύπτει από το άρθρο 63, σελίδα 67, όπου η δυνατότητα προκαταβολών ανέρχεται στο 50%. Η σελίδα, ε, στη σελίδα 59, άρθρο 49. Προβλέπε, ε, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο ορισμός της μεγάλης επιχείρησης γιατί θα είναι πολύ σημαντικός ο ορισμός αυτός. Ανάλογα με τη διευκρίνηση θα δοθεί η ενίσχυση του αλείς. Αν είναι ανεπαρκής η διευκρίνηση μπορούν να στερηθούν τη βοήθεια αλείς που επίσης θα πρέπει να περιληφθούν κάποιες συστάσεις στα κοινοτικά έγγραφα ώστε οι αλείς να έρθουν πιο κοντά στους καταναλωτές. Αναφέρεται στο άρθρο 41 η υποστήριξη δεν αφορά τις νέες ηχθιόσκαλες. Πώς όμως θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει ο ψαράς κοντά στον καταναλωτή αν δεν μπορεί να δημιουργήσει νέες ηχθιόσκαλες. Πολύ συχνά έχουμε το φαινόμενο να ψαρεύουν οι άνδρες ενώ οι γυναίκες να πουλούν τα ψάρια. Είναι το χαρακτηριστικό μιας οικογενειακής επιχείρησης. Πολύ συχνά και για γενές έχουμε στην Πολωνία το μοντέλο αυτό. Αν όμως ε, δεν υπάρχουν ε, σαφείς ε, μέτρα, σαφή μέτρα για την ενίσχυσή τους, δεν θα ενισχύσουμε τέτοιες οικογενειακές επιχειρήσεις. Αναφέρεται επίσης η δημιουργία νέων, νέων σημείων εκφορτώσεων θα πρέπει πραγματικά να δοθούν χρηματοδοτήσεις για, τέτοια νέα, νέες, για τέτοιες νέες εκφορτώσεις. Αλλιώς πώς έρθει κοντά στον καταναλωτή ο Αλίας. Άρθρο 61, σελίδα 65, αναφέρεται για να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων στα πλαίσια της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης θα πρέπει να καταλήξουμε σε μεγιστοποίηση της συμμετοχής ε, του τομέα Αλίας και της ιδεατοκαλλιέργειας στην αηφόρο ανάπτυξη το, της παράκτειας αλίας και της αλίας ανοιχτής θάλασσας. Οι αναφορές στην παράκτεια αλία, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, είναι πολλαπλές. Πολύ συχνά όμως αφορούν περισσότερο την ε, υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατάληψη του αλληλευτικού επαγγέλματος ή για αναπροσανατολισμό σε άλλα επαγγέλματα. Θα πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά περισσότερο την ελαχιστοποίηση της συμβολής του αλληλευτικού κλάδου στην οικονομία στις παράκτιες ζώνες και όχι στη μεγιστοποίησή του. Το νέο ταμείο ε, δεν προβλέπει εξυγχρονισμό των αλληλευτικών σκαφών, γιατί αναφέρεται ότι υποστηρίζεται εξυγχρονισμό του στόλου, προκειμένου όμως να μειωθεί η αλληλευτική προσπάθεια. Δυστυχώ, ε, δεν υπάρχει συνάφεια μεταξύ της πρόθεση του νομοθέτη και του, του διατακτικού. Γιατί πραγματικά είναι ελάχιστο το κέρδο των αλλιέων. Με έναν εξυγχρονισμό θα μπορέσουν να αλλιεύουν πιο αποτελεσματικά και να αλλιεύουν με τρόπο που θα προστατεύει το περιβάλλον. Δυστυχώ, ε, το, ε, το, το νέο ταμείο δεν προβλέπει τέτοια μέτρα και έτσι ε, δεν έχουμε δυνατότητα για νέε μεθόδου αλληλεία που θα προστατεύουν το περιβάλλον και θα προστατεύουν και του αλεί. Ο εξυγχρονισμό των αλληλευτικών στόλων, διατηρώντα το μέγεθο και την ισχύ του κινητήρα, δεν θα ε, συμβάλλει στην βελτίωση τη αλληλευτική προσπάθεια, αντίθετα θα βελτιώσει την κατάσταση των αλληλείων. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την αλληλεία γιατί δημιουργεί θέσει απασχόληση ε, επίσης δεν οδηγεί σε υπερβολική αλληλευτική προσπάθεια, αντίθετα συμβάλλει στην αηφόρο διαχείριση της αλίας και άρα στην αηφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας υπόψη την παρεμπίπτουσα αλία, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Να λάβουμε υπόψη και την υδατοκαλλιέργεια και την χρησιμοποίηση κάποιων μεθόδων εκτατικής αλίας, γιατί η Βαλτική είναι κλειστή θάλασσα. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες μεθόδους εκτατικής υδατοκαλλιέργειας όπως είναι η προστασία των τόπων ε, αναπαραγωγής, ο εμπλουτισμός με ελευτικά είδη ε, θαλάσσια, ο περιορισμός της ρήπασης της θάλασσας, γιατί όλοι αυτοί οι μέθοδοι θα ενισχύσουν την παραγωγή και θα μειώσουν τον ευτροφισμό. Ενώ οι μέθοδοι της έντατικής ε, ε, υδατοκαλλιέργειε, δηλαδή η χθιατροφή και η πάχυση των ψαριών θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του ευτροφισμού στη θάλασσα. Θα πρέπει τέτοιοι μέθοδοι να εφαρμοστούν στη Βαλτική, αλλά με πολύ μετριοπαθή τρόπο. Από αυτή την άποψη, το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Αλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστήμου του Τσέτσιν είναι έτοιμο για να εφαρμόσει εμπράκτος νέες μεθόδους και ε, να υλοποιήσει τους στόχους προς αυτή την κατεύθυνση. Η ζωή του αιλία είναι η καθημερινή επαφή με τη φύση σε ακραίες πολλές φορές συνθήκες. Οι Αλίες αποτελούν τμήμα του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ενδιαφέρονται περισσότερο από κανέναν, κανέναν άλλον για την καλή κατάσταση του αλληλευτικού αποθέματος και για τη βελτίωσή του. Αποτελούν τμήμα του οικοσυστήματος και το διαμορφώνουν. Προστατεύουν το περιβάλλον. Ας μην ξεχνούμε ότι επειδή ο αλληλεία είναι τμήμα του περιβάλλοντος ακριβώς, ε, έχει συμφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κατάσταση της αλληλεία στη Βαλτική χρήζει ιδιαίτερη μα και από μέρου των πολιτών, του κράτους αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ισχύον πρόγραμμα, στον άξονα 4, υπάρχουν κάποιε θετικέ διατάξει για του αλληλεί. Αλλά στην άπρο, ταμείο θάλασσα και αλληλεία, υπάρχουν πολύ λιγότερα τέτοια μέτρα. Αντίθετα, βλέπουμε μια επιδείνωση τη κατάσταση σε σχέση με τον τρέχοντα κανονισμό. Και οι δραστηριότητε στα πλαίσια του προγράμματο Αλία 2007-2013 θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν, να διασώσουν πολλέ θέσει εργασία. Α μην εξουδετερώσουμε λοιπόν τα, τα επιτεύγματα του προηγούμενου κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελικός ομιλητής είναι ο κύριος Μάρκος Νίγκε, σύμβουλο ε, σύμβουλος στην ομάδα PEW για το Ευρωπαϊκό Θαλάσσιο Πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να βρεθώ εδώ σήμερα. Θα αναφερθώ σύντομα στους λόγους γιατί οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ ενδιαφέρονται στις, ε, για τις επιχορηγήσεις ε, σχετικά με την αλία. Θα δούμε ορισμένα ζητήματα που απασχόλησαν το παρελθόν την κοινή αλληλευτική πολιτική και το Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας, τις προτάσεις και κάποιες συστάσεις μας για βελτίωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Αυτά τα νούμερα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ξέρετε, τα περισσότερα είδη ψαριών υπεραλλιεύονται. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Καντέκ, αλλά η πλεονάζουσα αλληλευτική δυνατότητα παραμένει το κύριο πρόβλημα που εντοπίζεται στην πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το έχουν αποδεχτεί και τα περισσότερα κράτη-μέλη εξάλλου. Επίσης, η αλληλευτικοί στόλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβαρύνουν τα ευθεία αποθέματα, αλλιεύοντας δύο ή τρεις φορές πάνω από το βιώσιμο επίπεδο και οι επιχορηγήσεις έχουν συνεισφέρει σε αυτό. Και το γεγονός αυτό, ότι οι επιχορηγήσεις δηλαδή συνεισφέρουν σε ε, αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας, και στην υπεραλίευση έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2002 στην ε, Παγκόσμια Διάσκεψη στο Johannesburg για την βιώσιμη ανάπτυξη. Μέλη του ΠΟΕ συναντήθηκαν στην Ντόχο για να διαπραγματευτούν τις επιχορηγήσεις για την αλία και αναγνώρισαν το γεγονό ότι δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα αυτό δεν είναι βέβαια κάτι καινούργιο, όμως γενικά την χάνει ευρύ αναγνώριση. Αρχή, θα αρχίσω ε, έτσι, κάνοντας μια γενική θεώρηση. Πού πηγαίνουν τα μεγαλύτερα κονδύλια, ποιο είναι το μοτίβο των ε, δαπανών. Οι περισσότερε επιχορηγήσεις πηγαίνουν σε ε, διαρθρωτικές ενέργειες στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελίας, περίπου ένα δισεκατομμύριο κάθε χρόνο για το ποσοστό προληπτική θνησιμότητας 46 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο πηγαίνουν στον έλεγχο και επιβολή του κανονισμού και αυτό είναι και ένα σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης των νυχθείων αποθεμάτων. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε όσους κανόνες θέλουμε και να είναι και πολύ καλοί αυτοί. Αν όμως δεν τους εφαρμόσουμε δεν μας βοηθούν καθόλου. Ο πίνακας εδώ σας δείχνει, εάν πάτε στο ποσοστό αλίας και κοιτάξετε τις δαπάνες και στο δεξί μέρος τα αποθέματα, θα δείτε ότι οι στόλοι που υπεραλλιεύουν τα συγκεκριμένα αποθέματα συνεχίζουν να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Ένα από τα μέλη αυτή εδώ τη Επιτροπής ερώτησε την ε, Επιτροπή για τις επιχορηγήσεις ε, αλίευσης ερυθρού τόνου και απάντησαν ότι ανάμεσα στο 2000 και το 2008 ο ευρωπαϊκό Τόλος έλαβε 33,5 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ευρωπαϊκά κονδύλια. Και όπως ξέρετε, ο ερυθρό τόνο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Εδώ λοιπόν θέλουμε να δείξουμε ότι ορισμένε από αυτές τις επιχορηγήσεις δεν βοηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, αρκετές φορές αναφέρθηκε το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις ε, βοηθούν κυρίως τις μικρές και μεσαίες ε, επιχειρήσεις και εδώ θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν μερικές αναλύσεις που δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης πηγαίνει στον αλλιευτικό στόλο, στα σκάφη δεν ε, καταλήγει απαραίτητα στις τσέπες των ε, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά στις μεγάλες. Εδώ θα δείτε ότι το, περισσότερο το μεγαλύτερο ποσοστό βοήθειας πηγαίνει στα σκάφη με ε, μέγεθος πάνω από 24 μέτρα. Ένα άλλο μικρότερο ποσοστό ανάμεσα στα 12 και 24 μέτρα και το μικρότερο ποσοστό σε σκάφη που είναι μικρότερο των 12 μέτρων. Θα δείτε ότι έγινε μια διάρθρωση των ε, χρηματοδοτήσεων των στόλων με χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Τα, ε, οι επιδοτήσεις αυτές ε, πήγαν σε ανακατασκευή των μεγαλύτερων σκαφών και η υποστήριξη των μικρών σκαφών είχε να κάνει κυρίως με διάλυσή τους. Εκεί λοιπόν πήγαν τα χρήματα των φορολογούμενων. Από, την, από την αλία μικρή κλίμακα στην βιομηχανική αλία. Αυτό δεν, είναι κατα... δεν θέλω να πω ότι είναι κατά αναγκή κακό, αλλά θέλω να το αναφέρω, ε, διότι οι επιχορηγήσει είναι προορισμένε για να βοηθήσουν τι μικρέ επιχειρήσει Και κοιτάξτε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Επίση, ε, να αναφερθώ σύντομα στο γεγονό ότι υπάρχουν αρκετέ επιχειρήσει, οι οποίε ήταν αναμεμειγμένε σε μεγάλες παραβάσει ε, όσον αφορά τη χρήση των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων είναι αρκετά δύσκολο να τηρήσουν αυτές οι επιχειρήσεις τους κανόνες. Δεν, δεν καταλαβαίνουν τα μειονεκτήματα και καταλήγουν να μην παίρνουν αυτές τις επιχορηγήσεις. Τώρα, όσον αφορά τις προτάσεις μας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας, μπορείτε να δείτε ότι υπήρξε μία αύξηση των ε, δαπανών για τα διαρθρωτικά μέτρα, υπήρχε λιγότερη για την συλλογή δεδομένων και για τον έλεγχο και την επιβολή. Αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι μια πραγματική μετάβαση από τα διαρθρωτικά μέτρα στη, στην συλλογή δεδομένων και στα ε, μέτρα ελέγχου. Οι δημόσιες ε, δαπάνες λοιπόν και δημόσιες επιχορηγήσεις πρέπει να ε, δοθούν σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι ανάγκη να καταβάλλετε τόσες μεγάλες προσπάθειες ελέγχου και σε γενικές γραμμές θεωρείται χρήσιμο την ε, διαχείριση της αλίας. Έπειτα, μέγιστα και ελάχιστα ποσοστά. Είναι καλό να εισαχθούν αυτά τα, τα ελάχιστα, το ελάχιστο ποσοστό δεδομένων για παράδειγμα. Όλα αυτά θα μας δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία για την μετάβαση της ε, χρηματοδότησης από τον ένα τομέα στον άλλο. Όπως ακούσαμε, ένα από μια από τις κυρίες ανησυχίες είναι η σύνδεση, η πιθανή σύνδεση ανάμεσα στην ε, αλλιευτική ικανότητα και στις επιχορηγήσεις. Ο... Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας ε, έχει κάποια μέτρα για τον ε, έλεγχο, για τον εξυγχρονισμό των αλλιευτικών σκαφών. Δεν περιλαμβάνει όμως την αντικατάσταση των κινητήρων σε αυτά τα σκάφη. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι οποιαδήποτε βοήθεια προς αυτά τα σκάφη να γίνει υπό προϋποθέσεις μετά από αξιολόγηση των σκαφών αυτών. Δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστό τα κράτη-μέλη να μην εξετάζουν λεπτομερώς την ε, χωρητικότητα ενός σκάφους και να εισραίουν ευρωπαϊκά κονδύλια σε σκάφη τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Μετά, είμαστε επίσης υπέρ της ε, απαλυφής ε, μέτρων που είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Ακούσαμε το πρωί για διοικητικό φόρτο, για δυσκολία ελέγχου και εάν αυτά τα μέτρα απαλληφθούν, θα μειωθεί επίσης και η ανάγκη για έλεγχο. Εάν απλά υποστηρίξουμε τη συλλογή δεδομένων, την επιβολή ελέγχου και την έρευνα, πιστεύω ότι ο έλεγχος μπορεί να ελαχιστοποιηθεί και να προσανατολιστούμε στον εξυγχρονισμό των σκαφών σε άλλες δραστηριότητες. Βέβαια, ο έλεγχος ε, προς το πού πηγαίνουν τα κονδύλια πρέπει να αυξηθεί. Οι προσπάθειες να ελέγξουμε το πού πάνε αυτά τα κονδύλια. Πιστεύουμε ότι η χρηματοδότηση είναι ένα καλό εργαλείο για να δοθούν κίνητρα, από τα βασικότερα κίνητρα, Υπάρχει όμως... Υπάρχουν όμω προποθέσει για τα κράτη-μέλη. Αν τα κράτη-μέλη θέλουν να λάβουν αυτέ τι επιχορηγήσει, πρέπει επίση να υποστηρίξουν και του στόχου τη κοινή αλληλευτική πολιτική, χρησιμοποιώντα αυτά τα όργανα, εφαρμόζοντα τη συλλογή δεδομένων, εφαρμόζοντα του ελέγχου και τους, κανονισμ, ε, τους κανονισμούς. Εάν αποτύχουν να εφαρμόσουν αυ, ε, τους ε, κανονισμούς σε αυτούς τους τομείς, το να συνεχίσουμε να τους δίνουμε επιχορηγήσεις είναι κάτι που δεν είναι συνετό. Και ο βασικός, ο ε, βασική, ο βασικός κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει να υπάρχει τουλάχιστον ε, διάστημα ενός χρόνου ε, συμμόρφωσης πριν από την χρηματοδότηση. Αυτό για μας πρέπει να είναι η, είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση για, την, για τις επιχορηγήσεις και για την μείωση και την απαλυφή της πλεονάζουσας αλληλευτικής ικανότητας. Έπειτα, πιστεύουμε ότι το διάστημα συμμόρφωσης πρέπει να αυξηθεί σημαντικά. Τέλος, να σας πω δύο πράγματα για την ε, διαφάνεια και τη μετάδοση πληροφοριών. Είναι απολύτως σημαντικό οι πληροφορίες ε, για τους δικαιούχους, για το σκάφος που λαμβάνει την επιχορήγηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η πληροφορία, διότι αλλιώς είναι δύσκολο, ε, για να μην πω αδύνατο, να αξιολογήσουμε το καθεστώς αυτό δαπανών. Και η κοινωνία των πολιτών έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ε, στο να μάθει πώς ξοδεύονται αυτά τα χρήματα, πού πάνε υπό το ισχύον καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Και η πρόταση τη ε, Κομισιόν βελτιώνει αρκετά τα πράγματα, μπορώ να πω. Δίνει... Θα ήθελα να, δώσω, να... να παροτρύνω το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την διαδικασία διαφάνειας, διότι όποιο και είναι το αποτέλεσμα στο τέλος, σίγουρα είναι, ε, είναι αποδεκτό ότι όλοι ενδιαφερόμαστε ε, να διοχετεύουμε τα κονδύλια στα, τι σωστέ δραστηριότητε, να εντοπίζουμε τα προβλήματα και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το σύστημα. Είναι απόλυτα λοιπόν σημαντικό αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες, οι πληροφορίες για το πώς ξοδεύονται τα κονδύλια. Και συνοψίζοντας τέλο. οι κύριες βασικές προτάσεις που θέλουμε να δώσουμε στο Κοινοβούλιο είναι η μετάβαση τη βοήθεια περισσότερο στην, ε, στο, στην συλλογή δεδομένων και στον έλεγχο και στην επιβολή ελέγχου παρά στα σκάφη να, ε, η απαλυφή της πλεονάζωσης αλληλευτικής ικανότητας και η υποστήριξη και η ενίσχυση της ε, πολλαπλής συμμόρφωσης. Υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που υποστηρίζουν αυτέ τι θέσει. Νομίζω υπάρχουν και κάποιε εκθέσει από αυτού του οργανισμού με περισσότερε λεπτομέρειε στην είσοδο τη αίθουσα. Και κλείνοντα, σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να σα κάνω την παρουσίαση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κνίγκε. Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Κυρία Ρομπούστ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Είναι πάντα εξαιρετικά χρήσιμο να έχουμε εδώ εμπειρογνώμονες. Θα απευθυνθώ σε έναν ομιλητή όμως τώρα, διότι πραγματικά ε, θεωρώ πως αυτό ήταν ένα σημαντικό. Κύριε Φίσον, μιλήσατε για στενότερη συνεργασία. Πιστεύω πως δεν διαφωνούμε, δεν έχουμε και πολύ, διαφορετικές θέσεις. Οι κυρώσεις και οι κανόνες πρέπει να είναι αυστηροί και να ισχύουν για όλους. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της ισχύουσας αλληλευτικής πολιτικής είναι ο τρόπος ε, διαχείρισης και οι κυρώσεις. Οι ποινές, για παράδειγμα, στη Γερμανία είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι στην Ιταλία. Έχετε δίκιο σε αυτό που, λέτε στην, είπατε στην παρουσίασή σας, ότι οι αλληλείς που ε, συμμορφώνονται με, τις, ε, με τους κανόνες έχουν ε, το, θα έπρεπε να έχουν το μεγαλύτερο συμφέρον για μια καλύτερη νομοθεσία. Και αυτό είναι το συμφέρον μας κιόλας και το συμφέρον τους. Διότι φυσικά έχουμε πολλά να χάσουμε όταν παραβιάζονται οι κανόνες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή λύση. Έχω μια πρόταση και αυτή είναι. Εσείς λέτε να οι ποινές να απευθύνονται στους παραγωγούς. Όμως, εγώ διαφωνώ. Πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθούν οι οργανισμοί παραγωγής, αλλά και να επεξεργαστούν και να αποφασίσουν για τις ποσοστώσεις από κοινού. Έχουμε να κάνουμε με ευρωπαϊκή πολιτική, που ισχύει σε όλο τον τομέα της, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεξαιρέτως. Όταν εσείς λέτε ότι εγώ θέλω να διαχειριστώ τις ποσοστώσεις μου με το δικό μου τρόπο, έτσι ώστε να δώσω μια ε, λογική τιμή στα ψάρια που θέλω να πουλήσω, ή θέλω εγώ να καθορίσω το τι θα γίνει με τους εγώνους των ψαριών, με τα μικρά ψάρια ή με αυτά που πιάστηκαν κατά λάθο στα, στα δίχτυα. Πιστεύω όμως ότι χωρίς να έχω μιλήσει με αντιπροσώπους ε, των ε, παραγωγών, ότι έχει γίνει καλή δουλειά και πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό οι αλληλείς να αποφασίσουν μόνοι τους τι θα γίνει με τις ποσοστώσεις τους και πιστεύω ότι είναι αρκετά έξυπνο αυτό να διοργανωθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις. Τώρα, κύριε Καντέκ, δεν Πιστεύω πως δεν μπορώ να είμαι πιο σαφής. Ως ε, ο, οργανισμοί παραγωγών πιστεύω ότι εσείς έχετε την αρμοδιότητα να αποφασίσετε ποια πλοία θα διατηρήσετε, ποια θα ανανεώσετε και δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Καντέκ δεν μπορεί να να δει πώς θα διαχειριστούμε το θέμα με την πλεονάζουσα αλληλευτική δυνατότητα. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρούντι, Ο κύριος Γκρουμπάρτσικ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, τα θέματα που έθιξαν οι καλεσμένοι μας, τους οποίους ευχαριστώ θερμότατα, κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και αναφέρονται και στην έκθεσή μας για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Αναφέρθηκε το θέμα της, ε, των, της εναρμόνισης των κανόνων σε ό,τι αφορά την κατανομή των αλληλευτικών ποσοστώσεων και το θέμα της ε, νόμιμης εφαρμογής, ε, της νομότυπης εφαρμογής ε, και του σεβασμού και της συντήρησης των αλληλευτικών αποθεμάτων. Δυστυχώς έχουν γίνει πολλά λάθη. Υπάρχει ελλειπής συμμόρφωση με τους κανόνες, είναι εμφανής αυτές οι αδυναμίες και θα πρέπει να εξαλειφθούν αν θέλουμε μια γνήσια κοινή αλληλευτική πολιτική. Το ίδιο αφορά και την προστασία της παραδοσιακής ή μικρής κλίμακος αλίας και το θέμα της επαναπεριφερειοποίησης και το θέμα της αερασιτεχνικής αλίας και ο, δικό της, ο δικός αντίκτυπος είναι σημαντικός για, το, για τα ελληνευτικά υποθέματα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν μελέτες και για αυτό το θέμα, για την επιρροή της αερασιτεχνικής αλίας στα ελληνευτικά αποθέματα και στο οικοσύστημα. Δυστυχώς τέτοιες μελέτες δεν έχει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μερικές φορές τα κράτη-μέλη εκπονούν παρόμοιες μελέτες, αλλά τα πορίσματά τους δεν τα διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο καθηγητής Βαυζίνιακ μας μίλησε και για το θέμα της υδατοκαλλιέργειας που είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε, σε υδάτινες εξαμενές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μιλήσατε για τη χρησιμοποίηση περισσότερο, μεθόδο, ε, τη χρησιμοποίηση περισσότερο των μεθόδων της εκτατικής υδατοκαλλιέργειας. Μπορείτε να συγκεκριμενοποιήσετε τις προτάσεις, παρακαλώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκρομπάρτσικ. Ε, η κυρία Γέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Καντέκ, γιατί γενικώ ε, συνέταξε μία έκθεση που κατά τη γνώμη μου είναι και πολύ ενδιαφέρουσα ε, και αξιόλογη. Μπορώ να προσυπογράψω τα περισσότερα σημεία της, παρόλο που θα υποβάλω και γραπτός κάποιες τροπολογίες. Ε, ζητώ συγγνώμη γιατί δεν συγκράτησα το όνομα του τελευταίου μας ε, καλεσμένου. Μίλησε πάντως ε, για το σε ποιο βαθμό οι επιδοτήσεις συμβάλλουν στην υπεραλίευση. Διαφωνώ. Δεν πιστεύω ότι οι χορηγήσεις συμβάλλουν στην υπεραλίευση. Βέβαια διαφωνώ και για πολλά άλλα θέματα. Αλλά ερωτώ το τελευταίο καλεσμένο. Είπε ότι το κονδύλιο που προβλέπεται στο Ταμείο για την συγκέντρωση δεδομένων έλεγχο και επιθεωρήσεις, ε, το ποσό αυτό είναι επαρκές. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχει ένα αποθεματικό ενός δισεκατομμυρίου 47 εκατομμυρίων για άμεση διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ίσως ε, αυτά τα κονδύλια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Συμφωνείτε, γιατί με τα μέτρα αυτά θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε το στόχο της ε, αηφόρου αλίας και να αποφύγουμε την υπεραλίευση. Γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε και τον αλληλευτικό κλάδο και τις περιφέρειες ε, που χρειάζονται τέτοια στήριξη, γιατί πρόκειται για ένα τομέα που οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη είναι πολύ σημαντικό, ενώ αντίστοιχα τα μέτρα είναι ελάχιστα, πολύ μετριοπαθή και πολύ ανεπαρκή. Γιατί μερικές φορές επικρίνουμε δρυμύτατα και ανελαίητα ε, το ταμείο αυτό που είναι 6,5 δις, ενώ ε, δεν ε, έχουμε καμία επιφύλαξη προκειμένου να επιδεψιλεύουμε κονδύλια σε χρηματοπιστωτικού οργανισμού που μα οδήγησαν σε κρίση και σε καταστροφή. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό το 1 δισεκατομμύριο 47 εκατομμύρια. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ε, το κονδύλιο αυτό για τον έλεγχο ε, της παράνομης και άναρχης αλίας. Γιατί τα κράτη-μέλη σε μεγάλο ή μικρό βαθμό εφαρμόζουν κάποιες εγγύσεις για την αποφυγή, τον περιορισμό της παράνομης και άναρχης αλίας. Αναφερθήκατε σε ένα κονδύλιο, αλλά δεν μα μιλήσατε για τα μέτρα που θα πρέπει να, χρηματοδοτηθεί, να χρηματοδοτήσει. Βέβαια, φαντάζομαι ότι αυτό αποτελεί ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μια και εκπροσωπείται ένα μεγάλο φάσμα οικολογικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, με τι οποίε συμφωνώ σε πολλά αιτήματα, θα ήθελα να μα δώσετε και τη δική σα προσέγγιση για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Γκαρσία Γέρο, κυρία Φράγκα τώρα. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ε, πιστεύω ότι μία από τις βασικές αλλαγές που περιλαμβάνει ο νέος κανονισμός για το ΕΤΘΑ σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας έγκυται στο ότι ε, εξουδετερώνεται ο πρώτος άξονας που προέβλεπε ενισχύσεις στον αλληλευτικό στόλο. Καταργείται πια αυτός ο πρώτος άξονας και πιστεύω ότι η πρόταση αυτή σχετίζεται με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το βασικό κανονισμό Δηλαδή, καταργούνται οι ενισχύσεις προς τον στόλο και αντίθετα στο βασικό κανονισμό προτείνεται ένα μοντέλο διαχείρισης που είναι διαφορετικό από το ισχύον, που είναι ένα μοντέλο που στόχο έχει τη μείωση της αλληλευτικής ικανότητας μέσω της, ε, του συστήματος των ε, αλληλευτικών δικαιωμάτων. Οπότε, φτάνουμε σε ένα μοντέλο με μεταβιβάσιμες ε, αλληλευτικές άδειες. Εγώ βέβαια είμαι υπέρμαχος, θερμός υπέρμαχος αυτού του μέτρου των μεταβάσιμων αλληλευτικών αδειών. Δυστυχώς υπάρχουν αντιρρήσεις και στο Συμβούλιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σύστημα αυτό. Στο μέτρο λοιπόν θα πρέπει, στο βασικό κανονισμό θα πρέπει να προβλεφθούν κάποια μέτρα στο μέλλον για ενίσχυση του στόλου. Γιατί αν δεν αλλάξει ο προσανατολισμός, δεν πρόκειται να αλλάξει και το μοντέλο ενισχύσεων του στόλου. Δεν μπορούμε από τη μια να καταργούμε ένα τμήμα και το άλλο να μην υφίσταται καμία μεταβολή. Εγώ είπα από την πρώτη στιγμή ότι θα ήμουν υπέρ του περιορισμού ή κατάργησης των ενισχύσεων του στόχου 1, του άξονα 1, αρκεί το μοντέλο διαχείρισης να είναι ένα μοντέλο διαχείρισης που είναι προωθεί τη μείωση της ελευτική ικανότητας. Αλλιώς ε, η διατήρηση του αλληλευτικού, της αλληλευτικής ικανότητας είναι αδύνατη. Θα πρέπει να λάβουμε κάποιες αποφάσεις ε, ολικής. Εγώ ήμουν υπέρ της προσέγγισης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις ε, θα πρέπει να τροποποιηθεί το θέμα του άξονα 1. Συμφωνώ με τον εκπρόσωπο της PEW και διαφωνώ με τον εισηγητή μας, τον κύριο Καντέκ, γιατί το βασικό πρόβλημα του ευρωπαϊκού στόλου είναι η πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα. Αυτή μας οδήγησε στην υπεραλίευση. Ας μην ομφαλοσκοπούμε, ας μην απομονωνόμαστε από τον υπόλοιπο κόσμο, θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οπότε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα όλης αυτής της ανάλυσης. Γιατί αν δεν τροποποιηθεί το μοντέλο διαχείρισης, εγώ θα προτείνω επαναφορά των ενισχύσεων του άξονα 1. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του εκπροσώπου της PEW, υπάρχουν ενισχύσεις για την προσωρινή πάυση δραστηριότητας ή την διάλυση, αλλά με βάση το νέο μοντέλο διαχείρισης, που φαίνεται ότι ε, όλο και περισσότερο νερώνεται και αλλοιώνεται, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Θα ήθελα οι εκπρόσωποι του κλάδου να σχολιάσουν αυτό το ζήτημα που είναι κεφαλαιόδου σημασία κατά τη γνώμη μου. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα που σήμερα δεν ακούσαμε καθόλου, αλλά είναι πολύ σημαντικό και συνδέεται με την κατάργηση των ενισχύσεων ε, στο στόλο του έξονα 1 και σε ενισχύσεις για τη διάλυση των πλοίων. Ήταν κοινωνικές ενισχύσεις που στο παρελθόν συνδέονταν με την πάυση ελευτικής δραστηριότητας. Με εντυπωσιάζει που δεν ανέφερε κανένα εκπρόσωπο του κλάδου, γιατί αυτό το θέμα των κοινωνικών ενισχύσεων συνδεόταν στο, παρελθόν με τις ενισχύσει για την πάυση της ε, ε, ε, του ελευτικού επαγγέλματος. Ενώ κοπτόμαστε υποτίθεται για τα κοινωνικά δικαιώματα, τη στιγμή της αλήθειας ε, αποσιωπούμε ένα ζήτημα που κατά τη γνώμη μου έχει μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσουμε ε, τον πρώτο γύρο των Ευρωβουλευτών, ο κύριος Κούν. Äh, Θα είμαι σύντομος. Ε, όσον αφορά την, ε, την γαλλική παρουσίαση για τον Ατλαντικό, είναι μια τα αποθέματα του γάδου είναι σημαντικά. Ο γάδος είναι ένα από τα σημαντικότερα ψάρια, ψαρεύεται στον Βόρειο Ατλαντικό και το παράδειγμα με τον γάδο μας δείχνει πώς η περιφερειακή οργάνωση μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Αυτό μπορεί να, σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η Κομισιόν στη Βαλτική έγινε κάτι παρόμοιο με τις ρέγγες, όταν ο πληθυσμός της ρέγκας, η βιομάζα της ρέγκας είχε μειωθεί πάρα πολύ. Ψαρεύονταν 20.000 τόνοι ετησίως και μετά αυτό απαγορεύτηκε. Πήγαμε με τους ε, τοπικούς συνδέσμους αλλιών στην Επίτροπο και είπαμε ότι χρειαζόμαστε ένα ε, πολιτές σχέδιο διαχείρισης και τότε παροπλίστηκαν αλλιευτικά σκάφη. Έγινε περιφερειακή διαχείριση και καταφέραμε να αυξήσουμε τον πληθυσμό τη ε, Ρέγκα στη Βαλτική και με παρόμοιο τρόπο θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε και του ε, πληθυσμού στα από θέματα του Μπακαλιάρου. Χωρίς τις ε, και θα πρέπει να καταστεί σαφέ ότι εάν δεν παροπληστεί ο αλληλευτικός ε, στόλος δεν θα πάει ούτε ένα λεπτό ευρωπαϊκής επιχορήγησης σε αυτές σε αυτούς τους, ε, τις αλληλευτικές, αυτές τις επιχειρήσεις. Και παρεπιπτόντως να πω ότι οι ποσοστώσεις της Ρέγκα στη Βαλτική ανέβηκαν κατά 30% φέτος. και ορισμένες επιχειρήσεις έπρεπε να σταματήσουν να διακόψουν την λειτουργία τους. Και να επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας να μάθουμε ακριβώς τα νούμερα του αλληλευτικού στόλου σε κάθε κράτος μέλος της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κούν. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε η κυρία Φαμίνια να σχολιάσει, αλλά παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, όπως μόλις δημοσίευσε μια πρόταση, την πρόταση που θα έχετε αντιληφθεί, απλώς δύο λόγια για να αναγνωρίσουμε ότι άζουσα ικανότητα και οι άμεσες επιδοτήσεις στην πράσινη βίβλο έχουν προσδιοριστεί ως σοβαρά προβλήματα στον τομέα. δεν επέτρεψε να είναι βιώσιμη η κατάστασή του. Αυτό που εμεί επιθυμούμε είναι ακριβώ ένα βιώσιμο τομέα, ένα βιώσιμό κλάδος που να είναι ανταγωνιστικό χωρίς απευθεία επιδοτήσει. Γι' αυτό μετατοπίσαμε την ε, στήριξη από την πρόσβαση 1, από τον πρώτο άξονα μάλλον, στη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές της παράκτειας, στις περιοχές αλίευσης, Έχουμε διευρύνει αυτό το πεδίο και ελπίζουμε ότι οι αλληλείς αυτών των περιοχών θα μπορέσουν να συνεχίσουν να αλλιεύουν και να διαβιώνουν, να διαβιώνουν στις περιοχές αυτές, αναπτύσσοντας τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Αυτό είναι ένα μέρος μόνο της πρότασης, η οποία είναι ευρύτατη. Αυξήσαμε τη χρηματοδότηση για τον έλεγχο και για τη συλλογή δεδομένων και προσπαθούμε να προβλέψουμε και την αρισιμότητα που είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να δημιουργηθούν κίνητρα και για τους φορείς και για τα κράτη-μέλη. Όμως η πρόταση της Επιτροπής είναι επιτάπητος πλέον. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να μελετήσουν την πρόταση και να επεξεργαστούν προτάσεις. Ευχαριστούμε κύριε Φαμίνια. Θα δώσουμε τώρα την ευκαιρία στους καλεσμένους μας να απαντήσουν. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Καντέκ. Ε, με συγχωρείτε πολύ γρήγορα να απαντήσω στην κυρία Φράγκα και στην κυρία Ρόντουστ. Δεν είναι εδώ η κυρία Φράγκα, παρά δεν θέλει να ακούσει την απάντησή μου. Απλώς να πω ότι Σα καθησυχάζω, Λουκέ. Συχνά συναντιέμαι με τον κύριο Πίσω, ο οποίο είναι και κοινό Γάλλο και όπω θα διαπιστώσατε, συμμεριζόμαστε την ιδέα ότι η υλοποίηση των μεταβιβάσιμων αδειών αλλία δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο στα κονδύλια και στι αλληλευτικέ προσπάθειε. Διότι, όπω θα ξέρετε, μπορεί να υπάρχει συγκέντρωση αδειών. Μπορείτε να με ακούσετε, σα παρακαλώ. Κύριε Κνίγκε. Αυτό θα οδηγήσει σε συγκεντρώσει αδειών. Δηλαδή αυτό που αλλιεύουν 10 σκάφη σήμερα, 100 τόνους ας πούμε, 10 σκάφη 100 τόνους, θα είναι το ίδιο με ένα σκάφο αύριο. Ένα σκάφο 100 τόνοι. Δεν θα έχει καμία, κανένα αντίκτυπο στα αποθέματα αυτό. Η κυρία Φράγκα, και δυστυχώ. μίλησε για τον μικρό κόσμο της Γαλλίας. Όχι, δεν είναι μικρό κόσμο, σας διαβεβαιώνω. Πολλοί είναι οι συνάδελφοι από την Επιτροπή αυτή και από άλλε χώρε που συμμερίζονται τι απόψει μου, συμπεριλαμβανομένων των Ισπανών. Θα σα το πω τέλο πάντων. Κύριε Κνίγκε, θα δώσουμε έτσι καλώ το λόγο στου προσκεκλημένου. Απλώ σε αυτό που λέγατε προηγουμένω και που είπε και η κυρία Ρόντουστ. Μην μπερδεύουμε την αλληλευτική δυνατότητα και την ικανότητα. Άλλο πλεονάζουσα ε, η, ικανότητα και άλλο η υπεραλίευση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για λόγους που σας εξήγησα. Εδώ θα κινηθούμε σε σαφρά θεμέλια. Δύο διακριτά πράγματα είναι η υπεραλίευση και η αλληλευτική ικανότητα. Θα τα συζητήσουμε όμως και μετά. Γκαμπριέλ, σου πίνω πάλι το λόγο. Ευχαριστούμε κύριε Καντέκ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο με τους καλεσμένους μας. Φαντάζομαι όλοι θα θέλουν το λόγο. Παρακαλώ δύο λεπτά το πολύ ο καθένας για να διευκρινίσετε κάποια θέματα. Ξέρω ότι είναι σύντομος χρόνος, αλλά δεν έχουμε περισσότερο δυστυχώς. Θα σας δώσω το λόγο με τη σειρά που τον λάβατε στη δημόσια κρόση. Κύριε Ερμίδα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω απλώς ότι στην παρουσίαση που έκανα αναφέρθηκα σε προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με το ισχύον ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Έχει όμως και πλεονεκτήματα αυτό το Ταμείο Αλίας. Είχαμε 19 προγράμματα προσαρμογής του χρόνου για να προσαρμόσουμε την πλονάζουσα αλληλευτική ικανότητα στους υπάρχοντες αλληλευτικούς πόρους. Επίσης, ε, στηρίξαμε επενδύσεις ε, στα πλοία, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν αισθητά οι συνθήκες διαβίωσης στα πλοία και σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν οδήγησε σε υπεραλίευση, σε αύξηση της αλλιευτικής ικανότητας. Πρόκειται για ένα κλάδο που δημιουργεί πολλές θέσεις απασχόλησης και μάλιστα σε ζώνες που εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά και μόνο από την Ελία. Έχουμε σημαντικές επενδύσεις, γι' αυτό θα πρέπει ε, να συνεχιστούν αυτές οι ενισχύσεις γιατί πρόκειται για ένα κλάδο που έχει εξαγωγικό προσανατολισμό, πολύ σημαντικό. Επίσης πρόκειται για ένα τομέα που βρίσκεται σε ανασυγκρότηση. Οπότε η, τα κονδύλια του άξονα 1 και του ΕΤΑ θα πρέπει να διατηρηθούν για να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της αλληλευτικής προσπάθειας και της αλληλευτικής ικανότητας. Γιατί διαπιστώνουμε ότι πολλές επενδύσεις που γίνονται στο, στα πλοία μπορούν αρχικά να αυξήσουν την ικανότητα, αλλά δεν, αυξή, δεν αυξάνουν την αλληλευτική προσπάθεια. Απλώ αυξάνεται η ασφάλεια στο πλοίο. Και ε, δεν είμαστε κατά των ελέγχων, είμαστε υπέρ των ελέγχων και μάλιστα υπάρχουν έλεγχοι και σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Απλώς θα πρέπει να αποφύγουμε επικάλυψη ή πολλαπλασιασμό των ελέγχων που δεν θα εξυπηρετήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων του Ταμείου. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στόχο των κονδυλίων είναι να συνεχιστεί η αλληλεία, ιδιαίτερα η παράκτια αλληλεία και η οικονομική ζωή στι παράκτιες ζώνε. Αυτό επιθυμούμε και στην Ισπανία. Ο αλευτικός κλάδος, που είναι πολύ σημαντικός κλάδος της οικονομίας και που βρίσκεται κυρίως στις παράκτιες ζώνες, θέλουμε να συνεχίσει να επιβιώνει, να συνεχίσει τις ελευτικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και θα πρέπει το νέο ταμείο να μην φυστεί προσπαθειών, προκειμένου να συνεχιστεί η ανασυγκρότηση του αλευτικού κλάδου και να μπορούν να εξακολουθούν οι αλείς, να ζουν από την αλεία και να επιβιώνουν και οι παράκτιες περιοχές. Σας ευχαριστούμε. Σχεδόν τηρήσατε το δίλεπτο, κυρία Γιαντσέβα. Δεν θέλει ο κύριος Κούκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Στην συζήτηση ακούστηκε αρκετές φορές ότι το δημόσιο χρήμα θα πρέπει να θεωρείται και δημόσιο αγαθό και ως τέτοιο να χρησιμοποιείται. Νομίζω ότι η αυτάρκεια στην παραγωγή τροφίμων είναι πολύ σημαντική ε, από αυτή την άποψη του δημοσίου αγαθού. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Ένωση εξαρτάται υπερβολικά από τις εισαγωγές. Απέχει πόρο της ε, αυτάρκειας της επίσης Ακόμη και αν δίνουμε κονδύλια σε ιδιώτες για ιδιωτικές επενδύσεις, το ζητούμενο είναι ούτως ή άλλως ένα δημόσιο αγαθό. Η αυτάρκεια στην... Ε, και η επισητιστική ασφάλεια ο εκπρόσωπος των Πολωνών ε, αλλιών μα είπε ότι δεν είναι μόνο η φώκε πρόβλημα, αλλά και η κορμοράνη. Αυτό είναι αλήθεια. Η κορμοράνη είναι ένα πρόβλημα περισσότερο δεδομένο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα ήταν καλό λοιπόν να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα διαχείρισης για όλη την Ευρώπη και για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των κορμοράνων. Σας ευχαριστούμε κύριε Πισόν. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω σε ένα-δυο σχόλια που έγιναν σε σχέση με την εισήγησή μου. Ε, στην τελευταία διαφάνεια που αφορούσε τις τιμές για, το, για τη διάλυση, τα πριμ για τη διάλυση, θέλω να θέσω το θέμα του αν αξίζει να διατηρήσουμε αυτό το εργαλείο που εν μέρη μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε την πλεονάζουσα δυνατότητα ικανότητα μάλλον. Όπως είπε και η κυρία Φράγκα, στην τελευταία διαφάνεια βλέπαμε ότι στη Γαλλία κατά καιρού, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, είχαμε ένα τέτοιο θέμα με την πλεονάζουσα ικανότητα. Το πραγματικό πρόβλημα με την ισχύουσα ελευθερική πολιτική είναι ότι η επιτυχία της εξαρτάται από την καλή θέληση των διαφορών φορέων να την υλοποιήσουν ή να μην την υλοποιήσουν. Σε κάποιες περιοχές οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι περιφερειές ανέλαβαν την ευθύνη να υλοποιήσουν τα εργαλεία αυτά. Και πολλοί οργανισμοί έχουν κάνει τα απαραίτητα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τη ε, πλεονάζουσα ικανότητα. Αλλού όμω έχουν γίνει διαφορετικέ επιλογέ. Η πλεονάζουσα ικανότητα και παραμένει και συνεχίζει να δημιουργεί πρόβλημα. Εδώ δεν θέλουμε βεβαίω να έχουμε την ελαζονία ότι κάνουμε διδάγματα στου υπόλοιπου καθόλου, αλλά θα ήθελα να μιλήσω και για τι μεταβάσιμε άδειε. Το εργαλείο που θα οδηγούσε σε σωστή κατανομή των αδειών δυστυχώ δεν συνοδεύεται από μέτρα ή διαχειριστικά μέτρα που να είναι συλλογικά και διαφανή. Άρα δεν προσφέρει και τίποτε. Θεωρώ ότι δεν είναι αναγκαίο ένα τέτοιο εργαλείο. Με τι μεταβάσιμε άδειε λοιπόν. Δεν θα πρέπει να έχουμε υποχρεωτική εφαρμογή τέτοιου κανόνα σε όλη την Ευρώπη. Κάπου μπορεί να γίνουν διαφορετικέ επιλογέ. οι άδειε να ανατίθενται σε άτομα. Τώρα, μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να οργανωθούν σε ομάδε σε ενώσει. Αυτό είναι επιλογή. Δεν είναι αυτή η επιλογή των Γάλλων ψαράδων, αλλά και σε άλλα μέρη τη Ευρώπη δεν έχει γίνει αυτή η επιλογή. Αλλά τα σχετικά αποτελέσματα είναι τελείω αποδεκτά και να συμφωνήσω και μαζί σας. Είπαμε προηγουμένως για την Πράσινη Βίβλο ότι πολλά λέγονται για την πλεονάζουσα ικανότητα. Στην Πράσινη Βίβλο γίνεται και λόγο για την ανάγκη να ανατεθούν κάποια πράγματα σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό καθόλου δεν αναφέρεται στο υπάρχον σχέδιο κανονισμό, τόσο. Και αυτό είναι ένα θέμα. Είναι κρίμα. Και να κλείσω εδώ λέγοντα κάτι και για τον ε, εξεβονίμων για τον άμμο. Εδώ η το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε, δηλαδή αν θα εξετάσουμε τα πράγματα από τη σκοπιά του, τι τάσεις υπάρχουν ή αν θα τα εξετάσουμε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή, τα αποθέματα κάποιες φορές απειλούνται από την πλεονάζουσα δυνατότητα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Αλλά εάν δει κάποια στιγμή κανεί τι συνέβη τη στιγμή τη συνόδου του Γιωχάνεσμπουργκ. Μπορεί τότε να μην ίσχυε κάτι τέτοιο ένα συγκεκριμένο απόθεμα, αλλά να ισχύει μετά. Ευχαριστούμε ο κύριο Σεμιόλη. Παρακαλώ να παραμείνετε στα δύο λεπτά γιατί στι 12.30 ούτω ή θα πρέπει να διακόψουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να είχα ακούσει μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει ότι πέραν των κοντιλίων που αποδίδονται στου ελέγχου, κάτι θα προβλεφθεί και για την αριστεχνική αλία. Καταγράφω όμω για άλλη μια φορά την απροθυμία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο κράτου μέλου και περιφέρεια συμβαίνει τελικά και εδώ. Κάτι συγκεκριμένο τώρα για τις ε, άδειε εκμετάλλευσης στην Καμπανία. Έχει γίνει αυτή η δοκιμή για την ε, παράκτη αλληλεία μικρής κλίμακας με τα συγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης αλλά και για προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Το αποτέλεσμα πριν καν ξεκινήσουμε ήταν να ενδιαφερθούν για αυτή τη νέα δυνατότητα εμπορευόμενη η οποία ήταν πανίσχυρη. Για, τη μικρή, λοιπόν, για την παράκτια αλία μικρής κλίμακα, εάν συνεχίσουμε αυτήν και ακολουθήσουμε αυτή την τάση, θα επαναληφθεί κάτι που σήμερα γνωρίζουμε και από την περίπτωση του ε, ρυθρού τόνου. Οι 700.000 τόνοι τελικά δεν ε, είναι αντικείμενο διαχείρισης από του αλείς όπω παλιά, αλλά οι αλεί αυτοί είναι πλέον μισθωτοί και εργάζονται σε μεγάλα σκάφη. Τι ποσοστώσει αυτέ τι έχουν στα χέρια του Τη έχει στα χέρια τη μία και μόνο επιχείρηση, ένα εμπορευόμενο σε όλη την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν που ζητώ είναι να προστατεύσουμε την παράκτη αλία μικρή κλίμακα, να τη αφήσουμε την επιλογή, να χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτό όπω θεωρεί καταλληλότερο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Σιμιόλη. Ο κύριος Βαυζίνιακ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Ο κύριος Γκρουμπάρτσεκ μίλησε για την εκτατική υδατοκαλλιέργεια. Πολύ συχνά αναφερθήκατε στην υδατοκαλλιέργεια. Τι σημαίνει υδατοκαλλιέργεια? Σημαίνει καλλιέργεια της θάλασσας ουσιαστικά. Οπότε τέτοιο είδους καλλιέργεια εφαρμόζεται με δύο τρόπους, με εκτατικό ή με εντατικό. Ο εντατικός τρόπος καλλιέργεια. Ε, έχει στόχο την εκτροφή των ηχθείων και την πάχυση των ηχθείων και άλλων οργανισμών. Για παράδειγμα, έχουμε 15.000 ε, ε, πέστροφες που μπορούν να, θρέψουν μια πόλη 3.000 κατοίκων όταν είναι δεόντως παχές άλλες μεθόδους χρησιμοποιεί η εκτατική υδατοκαλλιέργεια που προστατεύει τους τόπους αναπαραγωγής, δημιουργεί τεχνητούς τόπους αναπαραγωγής, χρησιμοποιεί ένα είδους βιολογικό καθαρισμό μέσω των μυδιών στη Βαλτική για παράδειγμα. Ανάλογα με το μέγεθος της ε, υδάτινης λεκάνης και ανάλογα με το, σύστημα, ε, το οικοσύστημα και τα χαρακτηριστικά, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφόρους μεθόδους υδατοκαλλιέργειας. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε παντού τις ίδιες μεθόδους υδατοκαλλιέργειας. Δεν έχουμε μονοσήμαντε ενέργειες και μονοσήμαγε δράσει. Θα πρέπει να δούμε ακριβώ τι στόχο θέλουμε και ανάλογα με το στόχο μα να υιοθετήσουμε κατάλληλε μεθόδου. Ευχαριστώ. Muchas ευχαριστούμε κύριε Βαυζίνιακ. Τελευταίος ομιλητής, ε, ο κύριος Νίγκε. Ευχαριστώ πολύ. Τα κονδύλια μας είναι περιορισμένα και το ερώτημα το πού πρέπει να διατεθούν αυτά Υπάρχει. Το συμπέρασμα που βγάζω εγώ είναι ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε όλον τον τομέα της αλίας, αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε την κοινή πολιτική. Χρειαζόμαστε ε, συλλογή δεδομένων, χρειαζόμαστε ελέγχους και χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι όλοι κάνουν τη δουλειά τους καλά. Υπάρχουν και άλλα όμως μέτρα τα οποία ε, απευθύνονται σε ορισμένους ε, φορείς και είναι πιο ρηψοκίνδυνα. Πρέπει να διασφαλίσουμε Πρέπει να φροντίσουμε να μην γίνεται υπεραλίευση και να μην υπάρχουν ρηψοκίνδυνες αλλιευτικές πρακτικές. Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει υπεραλίευση χωρίς πλεονάζουσα αλλιευτική ικανότητα. Έχουμε, ο στόλος μας έχει χαμηλή, χαμηλό οικονομικό ε, κέρδος και έχουμε ενδείξεις για ορισμένες περιπτώσεις ε, πλεονάζουσας ικανότητας. Τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων πηγαίνουν σε σκάφη τα οποία έχουν αυτή την πλεονάζουσα ικανότητα ή ε, δημιουργούν απορρίψεις. Και είναι σημαντικό, γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχει έλεγχος, για να μην ξοδεύουμε στα τυφλά κονδύλια. Πρέπει να φροντίσουμε να εξισορροπήσουμε τον αλληλευτικό μα στόλο, να εξισορροπηθούν οι αλληλευτικες ευκαιριε ευκαιρίε. Ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχουν καταφέρει να κάνουν σωστές αξιολογήσεις και παρατηρούμε ότι υπάρχει αυξημένη πίεση στα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με αυτές τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι κάτι που είναι γραμμένο και έχουν συμφωνήσει και τα κράτη-μέλη εξάλλου για αυτές τις προϋποθέσεις και βλέπουμε ότι δεν τηρείται. Πρέπει λοιπόν να τηρείται μια ισορροπία, όπως είπα, και επίσης να δούμε και που θέλουμε να είμαστε στα επόμενα δύο χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε αναλόγως Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πολύ καλύτερο πλαίσιο στο οποίο να ε, λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση. Για Σας ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσουμε τη δημόσια κρόση θα ξαναδώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Καντέκ. Πριν λοιπόν καταλήξω ε, σε κάποια σύντομα συμπεράσματα, μια και επέστρεψε η Κάρμεν, θα της απαντήσω. Η Γαλλία δεν είναι μικροκόσμος. Γιατί δεν είμαι ο μόνος που έχω αυτή τη γνώμη. Πολλοί συνάδελφοι συμφωνούν μαζί μου και μάλιστα και μερικοί Ισπανοί. Ήθελα να το τονίσω τώρα που επέστρεψε η ε, Κάρμεν. Θα ήθελα να κατακλείδη να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους γιατί πραγματικά ήταν πολύ σημαντικές και ποιοτικέ μεστές οι παρουσιάσεις τους και θα ρίξουν φως και στις δικές μας εργασίες. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας θα πρέπει να αποτελέσει κυρίως ένα επανδυτικό εργαλείο στο μέλλον της ε, αλίας και της ε, το καλλιέργειε, δεν θα πρέπει ο επαναπροσανατολισμός των ελαιών να αποτελέσει ο καταγορία λίθο. Οι επενδύσει θα πρέπει να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του ελευτικού στόχου. Χρειαζόμαστε πιο επιλεκτικά, πιο σύγχρονα, πιο ε, φιλοπεριβαλλοντικά σκάφη, που να αυξάνουμε όμω την αλληλευτική ικανότητα. Επίση, θα καθορίσουμε το πλαίσιο ε, της ε, κοινοτικής για την επόμενη δεκαετία με του νέου κανονισμού. Βέβαια με τις εμπορικές ανταλλαγές και την επιστηστική εξάρτηση θα πρέπει να επενδύσουμε σε μια ανταγωνιστική και βιώσιμη και αλία και υδατοκαλλιέργεια. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήμουν λακωνικότατο. Σας ευχαριστούμε κύριε Καντέτ. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω και πάλι θερμά τους συμμετέχοντες. Κύριε Καντέκ, δεν είναι θέμα η πρόβλημα της Ισπανίας, είναι θέμα προσέγγισης που ε, εφαρμόζουμε για την αλία κάθε φορά. Και αυτό είναι το καλό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι έχουμε απόλυτη ελευθερία για συζήτηση, για συνεννόηση, μερικέ φορέ για διαφωνία, Άλλε φορέ Πάντω ήταν πολύ θετική αυτή η δημόσια ακρόαση, γιατί θα μα βοηθήσει να διαμορφώσουμε τη γνώμη μα, να αποκρισταλώσουμε τη γνώμη μα και να καταρτήσουμε και κάποιε τροπολογίε ανάλογα με την προσέγγιση που υιοθετεί ο καθένα. Ευχαριστώ θερμότατα τους καλεσμένους που ήρθαν και μας έκαναν τις παρουσιάσεις τους, αλλά να ευχαριστήσω και τους ευρωβουλευτές και τη γραμματεία και όπως πάντα και τις υπηρεσίες διερμηνίας. Σας ευχαριστούμε. Ραντεβού το απόγευμα στις 3 για τη συνέχιση της συνεδρίασης.